Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πάρα πολλά σημεία στη μέση διάταξη για σήμερα και αύριο. Και παρακαλώ να έχω την προσοχή σας, γιατί όπως έλεγα έχουμε πάρα πολλά σημεία να συζητήσουμε και δεν έχουμε τόσο χρόνο. Επομένως πρέπει να βάλουμε και λίγο αυστηρούς κανόνες για το πώς θα προχωρήσουμε σήμερα. Καταρχήν έχετε παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Θέλω απλώς ε, να σας αναφέρω ε, προσπαθούμε κάπως ε, να ρυθμίσουμε την ημερήσια διάταξη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα σημεία της ημερήσιας διάταξης σήμερα Πρέπει μέχρι τις 11.30 να έχουμε ολοκληρώσει τις συζητήσεις μας. Ε, περίπου μισή ώρα για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, μας μένει, γιατί στις 11.30 θα έρθει η Επίτροπος κυρία Χέντεγκαρντ. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό σημείο που θέλω να σας πω. Ε, μετά περνάμε στο σημείο που αφορά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ζητώ συγγνώμη που καθυστερούν τα πρακτικά, αλλά δεν είναι δικό μου σφάλμα. Θα έπρεπε να έρχονται λίγο πιο γρήγορα τα πρακτικά. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 ακαιρεότητα και διαφάνεια της αγοράς ενέργειας. Και παρακαλώ να έχουμε το νου μας την ώρα, να μην καθυστερήσουμε. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Χατζημαρκάκη. Και σας υπενθυμίζω, πρέπει να ολοκληρώσουμε μέσα σε μισή ώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σήμερα για άλλη μια φορά συζητάμε τις τροπολογίες ε, και τις συμβαστικές τροπολογίες και μπορώ να σας πω ότι μετά από πολύ καλή και πολύ στενή συνεργασία με το σκιώδη ηγητή κ. Γκέωργ Σβόμποντα, Σιμάνσκι και Τούρμες από 343 τροπολογίε ε, έχουμε φτάσει σε 33 συμβαστικέ τροπολογίε ε, και 300 ε, τροπολογίε. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Επίσης ήθελα να σας πω ότι ήταν πολύ καλή και η συνεννόησή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεννοηθήκαμε με τρεις ε, γενικές διευθύνσεις ε, που εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις μας και καταφέραμε να συνεννοηθούμε ε, γιατί είχαν και μια κοινή γραμμή και μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για τις συμβαστικές τροπολογίες που θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο. Ε, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση, θα ήθελα να πω το εξή. Το πεδίο εφαρμογή που έχουν ε, ε, μας έχει απασχολήσει στη συμβαστική τροπολογία 20 και 22 όπου κυρίως μιλάμε για τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Στις συμβαστικές λύσεις αναφέρονται και τα πιστοποιητικά εκπομπών και οι διαπραγματεύσεις ε, και τα παράγωγα προϊόντα για τα συμβόλαια εκπομπών εδώ υπάρχει η γενική βάση, αλλά δεν υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, μιλάμε για το φυσικό αέριο και για για τον ηλεκτρισμό, αλλά δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση όσον αφορά τα πιστοποιητικά. Ο οργανισμός ε, θα ενημερώνεται πλήρως, χωρίς να έχει όμως κάποιες αρμοδιότητες. Ο οργανισμός ε, Acer, ε, στην εργασία των ρυθμιστικών αρχών. Μετά μιλάμε για τη δικαιοδοσία. Τι ακριβώς έχουμε σχετικά με, την πληροφόρηση. Στην συμβαστική τροπολογία 12 υπάρχει αυτό. Μετά τι είναι προϊόντα χονδρικής στην αγορά ενέργεια, παραδείγματο χάρη συμβάσει για την παράδοση φυσικού αερίου και ρεύματο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι παράγωγα τα θέματα ε, της ε, ε, αποκάλυψης εσωτερικών πληροφοριών υπάρχουν στην Συμβαστική Τροπολογία 16, ιδιαίτερα για την αγορά φυσικού αερίου. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τον κανόνα de που υπάρχει στην Συμβαστική Τροπολογία 14 αυτός ο κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους μικρούς συμμετέχοντες στην αγορά ούτε για συναλλαγές κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο συναλλαγών για να μην επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τους μικρούς συμμετέχοντες. Συμφωνήσαμε ότι η Επιτροπή μέσω πράξεων κατεξουσιοδότηση θα μπορέσει να ορίσει το συγκεκριμένο κατόφλι για τον κανόνα de minimis. Αυτό το αφήνουμε να το ορίσουν οι πράξεις κατεξουσιοδότηση και έχουμε αφήσει και ένα ανοιχτό αριθμό όσον αφορά ε, ε, ε, τα γίγαβατ κατέτος αυτό θα, είναι κάτι που θα αποφασιστεί αργότερα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τα προϊόντα αυτά της αγοράς ενέργειας χονδρικής δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την αγορά για να είναι κάτω από το κατόφλι του κανόνα de minimis. Μετά για την υποβολή δεδομένων, ε, συμβαστική τροπολογία 20. Θα πρέπει να δίδονται οι πληροφορίε απευθεία στον οργανισμό ε, Acer και θα πρέπει να έχουμε ε, τις κατάλληλες δομές για την υποβολή δεδομένων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δομές που ήδη υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, η υποχρέωση υποβολής δεδομένων θα πρέπει ε, να περιορίζεται γιατί ε, τα δεδομένα θα μπορούν να μεταβιβάζονται άμεσα στον οργανισμό Acer. Δηλαδή ο οργανισμός λαμβάνει άμεσα τις πληροφορίες και θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπόλοιποι οργανισμοί, παραδείγματο χάρη ο οργανισμό, η ρυθμιστική αρχή στη Γερμανία, να ενημερώνεται παράλληλα ε, και να παραμείνει η δομή αυτή όσο δυνατόν πιο ελαφριά από τεχνικής πλευράς. Μετά στην συμβαστική τροπολογία 6 Μιλάμε για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που μεταβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές και εδώ έχουμε συμφωνήσει ότι ε, ε, στην Ευρώπη έχουμε τα καλύτερα, το καλύτερο επίπεδο δεδομένων όσον αφορά την προστασία των ε, δεδομένων και πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα που ισχύει με τον ΕΝΙΖΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών. Στην τροπολογία 15 μιλάμε για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση Υποστηρίζουμε τις πράξεις καταξιοδότηση υπό τον όρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι οι πράξεις καταξιοδότηση ε, έχουν την ε, εμπιστοσύνη μας και ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταβιβάζει τα κατάλληλα έγγραφα εγκαίρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίπτωση πράξεων κατεξουσιοδότηση θα πρέπει η Επιτροπή να φροντίζει να υπάρχει κατάλληλη διαφάνεια με τη συμμετοχή των καταλλήλων εμπειρογνωμόνων. Αυτά ε, ε, αρκούν για να δώσουμε εμείς και το Συμβούλιο τη συμφωνία μας. Ένα δύσκολο σημείο στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο ήταν ε, η καταγραφή των συμμετεχόντων στην αγορά και η αδειοδότηση των συμμετεχόντων στην αγορά. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει σύστημα αδειοδότησης, σε άλλα κράτη-μέλη όχι. Αυτό το συζητάμε στη Συμβαστική Τροπολογία 18 και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο καταγραφής των συμμετεχόντων, ε, ε, είτε απλό αρχείο είτε αρχείο αδειοδότησης ε, αν δεν υπάρχει ένα απλό αρχείο θα πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό ε, αρχείο καταγραφής των συμμετεχόντων. Και εδώ έχουμε αφήσει ανοιχτό το χρονικό περιθώριο, αλλά υπάρχει πίεση χρόνου και ξέρουμε ότι η Επιτροπή με πράξη κατά εξουσιοδότηση θα ορίσει το χρονικό περιθώριο για την καταγραφή. Την πιο ήπια μορφή δηλαδή. Περνώ στην εναρμόνιση των κυρώσεων τώρα εδώ υπάρχουν ε, πολλές διαφορές στα κράτη-μέλη και ε, αυτό μας απασχόλησε στη συμβαστική τροπολογία 9. Έχουμε ελάχιστα ε, επίπεδα κυρώσεων και αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανώτερες από το δεχόμενο κέρδος στο οποίο, στο οποίο απευθύνονται ως κυρώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η συμβαστική τροπολογία στην οποία καταλήξαμε και περνώ στα χρονικά ε, δεδομένα τροπολογίες 9 και 18, συμβαστικές τροπολογίες 9 και 18. Η Επιτροπή θα ήθελε στο πλαίσιο των πράξεων κατεξουσιοδότηση να ορίσει από πότε θα αρχίσουν να ισχύουν οι κυρώσεις και υπάρχει στο 2.01 ένα χ το χ είναι ο άγνωστος που θα δει από την Επιτροπή αργότερα για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Ένα τελευταίο σημείο, τα γραφεία συνδέσμου, τα liaison offices, υπήρχε μεγάλη πίεση από τη Σλοβενία σχετικά με το αν θέλουμε να έχουμε γραφεία συνδέσμου ή όχι. Οπουδήποτε έχουμε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, πάντοτε υπάρχει πίεση των κρατών μελών, του κράτου μέλους υποδοχής δηλαδή, να μην υπάρχουν γραφεία συνδέσμου. Και συμφωνήσαμε εδώ σε μια διατύπωση η οποία λέει ότι ο Οργανισμός συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών ενέργεια ε, θα έχει τους κατάλληλου πόρου στη Σλοβενία, πόρου προσωπικού και πόρου οικονομικού αντί γραφείου συνδέσμου να έχει τις κατάλληλες επαφές με τα, τους σημαντικούς τόπους διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για την πολύ εντατική συνεργασία. Συναντηθήκαμε τέσσερις φορές και είμαι ικανοποιημένο γιατί μπορώ να σας παρουσιάσω εδώ ένα πολύ καλό κείμενο και για τις συζητήσεις μας σήμερα και για την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ από τους επόμενους ομιλητές να προσέξουν να μην μακρηγορήσουν γιατί ήδη άρχισε να περιορίζεται ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή μας. Σκιώδης εισηγητές, ο κύριος Μπιουργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την ε, συνεργασία με τον εισηγητή Θεωρώ πως ε, και οι υπόλοιποι σκιώδεις ηγητές θα συμφωνήσουν ε, με το ότι ήταν πολύ καλή συνεργασία. Ελπίζω λοιπόν να συνεισφέρουμε στο ε, βελτίωση του σχεδίου Έκθεση εδώ πέρα. Είχαμε ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Κομισιόν. Βεβαίως το έργο μας ήταν εύκολο γιατί τα σημαντικότερα τα είχε ήδη κάνει ο, Οπότε καταφέραμε να έχουμε δύο συμβιβασμούς. Ο πρώτος αφορούσε το ίδιο το κείμενο, τις λεπτομέρειες, π.χ. το ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυτές τις παράλληλες εκθέσεις, αλλά ένας τέτοιος συμβιβασμός είναι και το πώς ορίζεται ε, πιο επακριβώς η εσωτερική πληροφόρηση. Και τα παραδείγματα που αναφέρονται εδώ πέρα θα συνεισφέρουν στην καλύτερη πρακτική εφαρμογή. το άλλο είδος ε, συμβιβασμών αφορούσε εκείνους τους που πάνε πέρα από το αρχικό πεδίο της πρότασης, δηλαδή αυτά που αφορούν το διοξείο του άνθρακα, εναρμόνιση των αδειών και εναρμόνιση των κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου την πραγματικότητα. Π.χ. όσον αφορά τις άδειες θεωρώ πως το σύστημα καταγραφής είναι ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός που μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το νομοθέτημα αυτό και να έχουμε και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως αυτή ήταν η δυνατότητα ε, να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία συνοψίζοντας θεωρώ πως καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό μέσω της συνεργασίας και μέσω των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο θα επιτύχουμε να τεθούν ενισχύτως το στομότερο δυνατόν αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Ριέρα Ματουρέλ που εκπροσωπεί τον κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Φόποντα, ο εισηγητής μας, ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να παρευρεθεί η σημερινή συνεδρίαση. Μου ζήτησε δε. Να σας πω ότι η ομάδα μας είναι πλούς ικανοποιημένη από τις εργασίες του εισηγητή, διότι έδειξε ένα πνεύμα συνεργασίας και Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Για τις τροπολογίες ήθελα να σας πω μόνο ότι πέρα από την πολύ καλή παρουσίαση του κυρίου Χατζημαρκάκη θα υποστηρίξουμε και εμείς τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύουμε ότι υπάρχει ομοθυμία στο Κοινοβούλιο και άρα θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική μας θέση ενώπιον του Συμβουλίου στον ε, επικείμενο τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Τζιμάνσκι. Ευχαριστώ. Ε, είχαμε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις ε, εισηγητές ε, και καταλήξαμε σε συμβαστικές τροπολογίες σχεδόν για όλα μας τα προβλήματα. Υπάρχουν βεβαίως πιο ακαθόδη ζητήματα στην ενεργειακή αγορά ε, και τέλος πάντων τελικά έχουμε μια ευρεία συνένεση. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω δύο θεμελιώδη για τους συντηρητικού ζητήματα. Πρώτον, δεδομένα. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, δια, διαφανή διαχείριση των απαιτούμενων δεδομένων και χρειαζόμαστε το μέγιστο δυνατό ε, βαθμό αξιοπιστίας ε, και χρειαζόμαστε την κατάλληλη τεχνική υποδομή για την διαχείριση των δεδομένων. επίση για τη δημοσίευση αυτών χρειαζόμαστε ε, σαφείς κανόνες. Τώρα για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω. Ε, δεν αφορά μέσα βέβαια το, το κοινοβούλιο αυτό το θέμα που σχολιάζω. Χρειαζόμαστε πάντως ένα σαφέστατο ορισμό Χρειάζεται συνεργασία από πλευρά του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να εκπροσωπούνται και οι φορεί τη αγορά. Θεωρούμε ότι η διατύπωση του ορισμού είναι καλή και άρα θα υποστηρίξουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση, τη θέση δηλαδή του Κοινοβουλίου, που υποστηρίζει και ο εισηγητή μα, ο κ. Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Κλοντ Τούρμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Χατζημαρκάκη, τον εισηγητή, ο οποίος βεβαίως ε, μας ε, και όλους και βεβαίως δεν έκανε αυτό το οποίο έχουμε συνήθως, δηλαδή να δεχτεί πίεση από εθνικές ε, κυβερνήσεις και να δεχτεί τελείως εθνικά επιχειρήματα. Το αρνήθηκε αυτό και είναι προς του ε, και δείχνει μια ευρωπαϊκή σκέψη. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε χάρη στον κύριο Γιούρκης ήταν να κλείσουμε πιθανά παραθυράκια στην νομοθεσία αυτή και ελπίζω αύριο να έχουμε συνέπεια και στην ψηφοφορία μας. Έχουμε λοιπόν την 188, 182 και την 86. Και ειδικά η 88 και η 66 των κυρίων Ρόιλ, πρόκειται για τις τροπολογίες του ΕΛΚ, είναι τροπολογίες που πάνε κατά της συμβαστικής μας λύσης και ελπίζω να μην ξανανοίξουμε αύριο παραθυράκια που προσπαθούμε να, προσπαθήσαμε να κλείσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις. Επίσης, ε, σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σαφές πως η αγορά διοξιδίου του άνθρακα συνδέεται με την τιμή του ηλεκτρισμού, τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρισμού και ελπίζω η Acer να το ε, παρακολουθεί. Και βεβαίως έχει έτσι αρκετή εξουσία η Acer. Θα καταθέσουμε μια τροπολογία ως πράσινη και δίδεται έτσι ρόλος και στην περιφερειακή συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, ειδικά καθώς η αγορά θα γίνει πιο περιφερειακή και κάτω από τους εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Acer πρέπει να αναφέρουμε ειδικά την σημασία της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών αρχών. Π.χ. η, π.χ. η αγορά Γερμανίας, Γαλλίας, Μπενελούξ, η πενταμε... αυτή αγορά. Και αυτό θα πρέπει ε, να βοηθήσει να σταματήσουμε εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και να έχουμε και περισσότερη διαφάνεια και ρευστότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις αγορές ηλεκτρισμού και αερίου και έτσι ελπίζουμε πως αυτό το οποίο έχουμε δηλαδή να δώσουμε περισσότερες εξουσίες ε, στην Acer και περισσότερες ε, διμερείς και έξω χρηματιστηριακές συναλλαγές να έρθουν εντός του χρηματιστηρίου να μπορέσουμε να το περάσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίρεκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, αλλά ο κίνδυνος κερδοσκοπίας στις αγορές αυτές πρέπει να περιοριστεί. Πρώτον, με, την, με τον περιορισμό της απαιτούμενης περίοδου για τη μεταβίβαση των πληροφοριών, για να μην υπάρξει κατάχρηση από τους φορείς αγοράς. Δεύτερον, τα επιστημονικά ιδρύματα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της Λιουμπλιάνα, του οργανισμού δηλαδή, για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια τρίτων. Η ε, εξαγορά της αποθηκευμένης ενέργειας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Taip pat noriu prisidėti prie visų padėkų. Ο κύριο ε, Μπατσίτη, ε, ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ευχαριστήσω τον συγητή για ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχει συνταχθεί εδώ και δύο χρόνια, το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε ορίσει. Η ολοκλήρωση της κοινή αγοράς απαιτεί ένα κοινό σύστημα για την παρακολούθηση και έλεγχό της και θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα πρέπει να επιλέξει κεντρική αγορά αερίου για να μπορέσουμε να έχουμε διαφάνεια τιμών για τους ε, καταναλωτές. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα εξαρτηθεί από το πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την αγορά ενέργειας. Η κατάχρηση και οι παράνομες δραστηριότητες ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν αν έχουμε ένα κοινό σύστημα ποινών, ένα ενιαίο σύστημα ποινών. Αναφέρθηκε πως ε, κάθε κρατος μέλος θα ορίσει ελάχιστες προδιαγραφές για τις ε, ποινές. Στην αρχική φάση μπορεί να μοιάζει κάτι τέτοιο ε, λογικό, αλλά μακροπρόθεσμα η υπηρεσία αυτή, η Acer, θα πρέπει να έχει ευρύτερη εντολή για να καθορίζει τις ποινές. Όπως συμβαίνει τώρα με την ε, Κομισιόν που ορίζει ποινές για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Οπότε σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές στο πολύ σημαντικό αυτό έργο. Ε, Μαρινκιέβιτς. przewodniczący. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την ε, έκθεση. Καταλήξαμε σε συμβαστικές ε, προτάσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να αλλοιώσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απελευθέρωση των αγορών και των ενεργειακών υποδομών. Οπότε, με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζουμε το συνελικό πακέτο μέτρων και ενισχύουμε την ε, διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά και προωθούμε την ολοκλήρωση. Η εναρμόνιση των εθνικών ενεργειακών αγορών και των, της εθνικής νομοθεσίας συμβάλλουν στην επίτευξη του ίδιου στόχου. Τώρα θα πρέπει να άρουμε τους τελευταίους φραγμούς ε, και νομίζω ότι πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να μην υπάρχουν προσκόμματα κατά τη θέση σε εμπορία και ε, στις αγορές ε, χοντρικής ε, για την ενέργεια Τίποτα δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης θα πρέπει να είναι ευκολότερο στις διασυνοριακές συναλλαγές να εντοπίζουμε τις παραβιάσεις της νομοθεσίας. Τέλος, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο μητρό Μόνο έτσι θα επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τις ε, ρυθμιστικές ε, αρχές και τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να κατοχυρώσουν και την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Εξού και τροπολογίες για την πιστοποίηση των ρυθμιστικών αρχών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Ουγγρική Προεδρία για την επιτυχία στο φάκελο αυτό. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο πολύ γρήγορα στην Επιτροπή, αν το επιθυμείτε. Κύριε Μπέρναρτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς από την πλευρά μα ευχαριστούμε τον εισηγητή και του σκιώδει εισηγητέ για τη δουλειά που έγινε. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Θα εξετάσουμε και τις λεπτομέρειες των συμβιβαστικών τροπολογιών, αλλά επί της αρχής δεν βλέπω κάποια μείζωνα δυσκολία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τον Ιούνιο στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Ωραία. Καλά ακούγονται και αυτά που μας είπε η Επιτροπή. Ο κ. Χατζημαρκάκης. Ε, υπάρχουν διαπραγματεύσει ε, με το Συμβούλιο ε, στις οποίες ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια σημεία αλλά γενικά οι πολιτικές ομάδες νομίζω ότι μπορούν να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι κινούμεθα προ μια κοινή κατεύθυνση και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί μα έχει προετοιμάσει πολύ καλά το έδαφο και εμεί βέβαια ω Κοινοβούλιο όπω πάντοτε βελτιώσαμε αυτό που μα είχε ετοιμάσει η Επιτροπή. Ωραία. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, λέει ο πρόεδρο. Ε, ενίοτε υπάρχουν προβλήματα, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν τίποτα. Αύριο ψηφίζουμε για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ γιατί ολοκληρώσαμε μέσα σε μισή ώρα αυτό το σημείο, χωρίς να σας πιέσω. Και περνάμε στο σημείο 6, έλεγχος των κινδύνων που συνδέονται με τα μείζωνα ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες. Ένα. Σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια και μετά θα ασχοληθώ ει βάθο ε, με το θέμα. Η οδηγία σε βέζο για τη διαχείριση των βασικών κινδύνων των επικίνδυνων ε, ουσίων έχει ως στόχο την πρόληψη ε, ατυχημάτων που ενέχονται επικίνδυνε ουσίε, τον περιορισμό των συνεπειών και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον και την υιοθέτηση προληπτικών πετούμενων μέτρων. Τώρα για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Ενδιαφέρεται κυρίω η χημική βιομηχανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδραξε την ευκαιρία της αναθεώρησης της οδηγίας που απαιτεί το επειδή θα υιοθετηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση, ε, την ετικετοθεσία ε, και των ουσιών καθώς και των παρασκευασμάτων. Έδραξε λοιπόν την ευκαιρία της αναθεώρησης για να τροποποιήσει αυτή την οδηγία που δεν είχε υποστεί καμία τροποποίηση από την υιοθέτηση της και μετά. Προτείνεται το εξή απλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα προβούν σε μια απλή εξοραϊστική δράση. Ε, θα βάψουμε μόνο το σπίτι ή θα κάνουμε κάτι ε, για να αποτρέψουμε τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί από το 1996 και μετά που έχουν καταστροφικές συνέπειες και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχουν βασικοί κίνδυνοι για την υγεία. Τροποποιούνται οι κατηγορίες. Η παλιά κατηγορία πολύ τοξικές ε, τώρα έχει αντικατασταθεί με την πρώτη κατηγορία, οξία, τοξικότητα κτλ. Ε, υπάρχουν υποκατηγορίε ε, πολύ ειδικέ ε, που βάσει του κανονισμού CLP που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και αντικαθιστούν τι γενικότερε παλαιότερε κατηγορίε που αντιστοιχούν στι εκρηκτικέ αυτοαναφλεγόμενες ουσίες και δεν έχει γίνει άλλη ουσιαστική τροποποίηση. Τώρα, έχουμε νέους κανόνες για την πρόσβαση για το κοινό, νέοι κανόνες για την ασφάλεια, πρόσβαση προσφυγή στη δικαιοσύνη και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προφανώ, οι ανακοινωθήσεις, ε, αλλαγές, δεν προκαλούν την ίδια ε, εντύπωση και αντίδραση σε όλους. Είδατε τι έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τώρα, ε, η για τις εταιρείε ε, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλά για τη χημική βιομηχανία θεωρούμε ότι θα σημειωθεί αύξηση πάνω του 10%. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τώρα θεωρούμε ότι παρότι είναι σωστή η γενική κατεύθυνση, ε, υστερεί το κείμενο για βασικά ε, θέματα. Ποιο είναι το ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Θα ε, κοιτάζουμε να, να περνάει το τρένο ή θα ανέβουμε πάνω και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τους κανόνες για την ασφάλεια. Ε, και ό,τι σχετίζεται με την βιομηχανία. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και περιμένω τη συνεργασία σα. Ε, με την ιδιότητα του συγητή θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσεις. Πρώτον, γενικέ, Προτείνει το κείμενο διάφορες δυνατότητες παρέκκλησης, ε, δυνατότητες δηλαδή παράκαμψης ε, των αρχών πρόληψης ε, που προτείνει η οδηγία. Αυτό είναι προβληματικό. Δεύτερον, τα δικαιώματα που εκχωρούνται στους μισθωτούς και στα όργανα εκπροσώπησής τους καθώς και στις ενώσεις τους μειώνονται σε αμεληταία ποσά. αντίθετα, μιλάμε για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το κοινό. Υπάρχουν δύο πλήρη άρθρα. Αντίθετα, σχεδόν δεν υπάρχει καμία αναφορά στο προσωπικό των επιχειρήσεων και ούτως ή άλλως ό,τι όποια αναφορά υπάρχει συγκεντρώνεται μέσα σε ένα άρθρο. Ε, και δεν υπάρχει και τίποτα σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και το ρόλο τους. Αντίθετα, στο άρθρο 20 που μιλάμε για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εκεί δίνεται έμφαση για την απαιτούμενη πρόσβαση για το κοινό και οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση δρά υπέρ του περιβάλλοντος ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επαρκέ συμφέρον ώστε να δράσει. Αντίθετα όμως οι εκπροσωπευτικές συνδικαλιστικές ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν ε, το ίδιο αυτονόητο δικαίωμα να παρέμβουν. Πρέπει να διορθώσουμε λοιπόν αυτή τη θέση των μισθωτών όπως φαίνεται στην οδηγία. Για τα παραρτήματα τώρα ε, δεν αναφέρεται καθόλου ο κίνδυνος που σχετίζεται με την απώλεια ελέγχου βιομηχανικών δραστηριοτήτων κινδύνου λόγω υπεργολαβίας. Ε, όμως σε πολλούς φακέλους η υπεργολαβία ακριβώς ήταν που δημιουργούσε τα προβλήματα. στην Τουλούζη η περίπτωση Αζεντεφ κατέδειξε η δικαιοσύνη είναι παραδείγματο χάρη, ότι η επιλογή τη υπεργολαβία και οι δυσκολίε που υπήρχαν για την μεταφορά τη τεχνογνωσία οδήγησε σε, εκατοντάδες, σε δεκάδε θανάτου, σε απώλεια στέγη για εκατοντάδε κατοίκου κτλ. Ε, η οδηγία δεν ανα... Ε, μέσα στην οδηγία δεν αναρωτιόμαστε επίση για την εμπορική αυτή σχέση που πρέπει να υπάρχει για την πρόληψη των κινδύνων. Μόνο στο άρθρο 11.4 προβλέπεται διαβούλευση με του υπεργολάβου. Μια απλή διαβούλευση δηλαδή δεν επαρκεί αυτό για να διαχειριστούμε τέτοιου είδου προβλήματα. Επίση, άλλα προβλήματα τίθενται στο σχέδιο μέσα ο συντονισμός παραδείγματος χάρη τη δράση των αρμοδίων αρχών. Ωραία. Τι γίνεται όμω με τα πρακτικά που θα συντάσσουν οι ελεγκτικέ αρχέ σχετικά με το εργατικό δίκαιο. Επίσης αναφερόμαστε στα επικουρικά υλικά μέσα, τα οποία όμως είναι ατελή και δεν προβάλλονται επαρκώς. Ε, ούτε και έχουμε αναφορά για την αποκόμιση διδαγμάτων από τα ε, παλιά ατυχήματα που έχουν ήδη σημειωθεί επίσης στην ακρόαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, συζητήθηκαν ε, βασικά προβλήματα όπως οι φυσικές καταστροφές και οι μεταφορές επικινδύνων ε, ουσιών. Η έσχατη καταστροφή της Φουκουσίμα έδειξε εξάλλου ότι τον λαμβάνουμε υπόψη μόνο τους τεχνολογικούς κινδύνους δεν επαρκεί και δεν συνιστά πρόσφορη πολιτική για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και του προσωπικού και του παρακειμένου πληθυσμού και άρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη θέση για τι φυσικέ καταστροφέ τώρα για τη μεταφορά των επικινδύνων ουσιών. Ε, υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι για του οποίου πρέπει σαφέστα να υπάρχει αναφορά στην ε, οδηγία σε Βέζο 3 για τη μεταφορά των επικινδύνων ουσιών. Πρώτον, όλοι το γνωρίζουν, α μην κάνουμε ότι είναι μυστικό η μεταφορά των επικινδύνων ουσιών ε, χρησιμοποιείται από διαφόρου ε, βιομηχανου που θέλουν να είναι κερδοφόροι και όχι υπεύθυνοι ενώπιον ε, τη κοινή για να αυξήσουν τα βασικά του αποθέματα παρακάμπτοντα έτσι κανονισμού. Ε, για την ασφάλεια σχετικά με τα ανώτατα κατόφλια για την αποθήκευση. Άρα είναι λογικό η μεταφορά των επικινδύνων ουσιών ε, που συνδέεται με αυτή την εξωτερήκευση να μετακυλίεται στα βασικά αποθέματα των επιχειρήσεων αυτών ε, και να χρησιμοποιείται για να παρακαμφθεί η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Έτσι, ε, μόνο αναθεωρήσουμε αυτή τη διάταξη θα μπορέσουμε να καταστήσουμε πιο ασφαλή την οδική κυρίως μεταφορά των επικινδύνων ουσιών γιατί οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να προαγάγουμε παράγουμε και την πολυτροπική, διατροπική μεταφορά των επικίνδυνων ουσιών στη συνέχεια. Ιδού λοιπόν ε, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να ε, συμμετάσχουμε όλοι στη συζήτηση. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και θα τις λάβουμε υπόψη εάν ε, ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Αυξημένη ασφάλεια δηλαδή για όλους, για το προσωπικό, για τις επιχειρήσεις, για τον πληθυσμό, για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Okay. Dann darf ich als ersten Herrn Δίνω το λόγο στον κύριο Μεζάρος καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Σκιώδης εισηγητής από το ΕΛΚ θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνο ε, σοβαρών ατυχημάτων ε, σε θέματα που συζητούμε με σοβαρέ συνέπειε. Ε, και γνωρίζουμε ότι με την καταστροφή με την ηλί στην Ουγγαρία είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα όπως και στην Τουλούζη επίσης. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλε οι επιπτώσεις για το περιβάλλον από τέτοια ατυχήματα. Γι' αυτό χρειάζεται ο εξυγχρονισμό της οδηγίας σε 2 και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η οδηγία αυτή αφορά περίπου 10.000 επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε ε, να μειώσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων που έχουν σχέση με χημικές ουσίες. Αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας. Από τότε που εγκρίθηκε η οδηγία έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις. Θέλουμε στο μέλλον να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και γι' αυτό χρειάζεται ο εξυγχρονισμός συγκεκριμένων μέτρων και πρέπει να πω ότι η τωρινή οδηγία σε ΒΕΖΟ 2 είναι αποτελεσματική και οι διαρθρώσεις και τα διάφορα μέτρα τα οποία προβλέπονται ε, ε, δεν χρειάζονται αλλαγή. Ο κύριος λόγος ε, για τον οποίο χρειάζεται τροποποίηση είναι το παράρτημα. Το παράρτημα χρειάζεται εξυγχρονισμό και θα πρέπει η ταξινόμηση σε κατηγορίες να γίνει με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στους σημερινούς κινδύνους και θα πρέπει να καθορίζονται ε, τα κατόφλια που θα ισχύουν ε, για τη δήλωση των ε, στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να μην ξεπερνιέται το κατόφλι του 3 5% για να ορίζεται ε, αν κάποια ουσία είναι ε, ε, σε ποια κατηγορία εντάσσεται κάθε ουσία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οδηγίας αυτό που αφορά την ταξινόμηση και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση με το σωστό τρόπο. Το περιεχόμενο της τροπολογίας 7 είναι σημαντικό όσον αφορά τα κριτήρια και θα πρέπει να μπει στο νέο νομοθετικό κείμενο. όσον αφορά την πληροφόρηση θα πρέπει οι πιο σημαντικές πληροφορίες να δημοσιοποιούνται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν τι είναι ε, κατάλληλο ε, να κοινοποιείται και τι όχι. Εδώ χρειάζεται κάποια ενερμόνιση ε, του τρόπου με τον οποίο θα δημοσιοποιούνται τα αποτέλεσμα των ερευνών και κατά αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιήσουμε και το διοικητικό άχθος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χίτσκο. Αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε. Ουλσκοκ, η κυρία Ουλσκοκ. Όχι, λάθος. Κυρία Γκριβάζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ενά, τον εισηγητή μας πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε σε μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην οδηγία. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ πρώτον με την πρόληψη. Θα πρέπει να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού τους κινδύνους που συνδέονται με την έκρηξη επικινδύνων ουσιών. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση των μισθωτών στο ίδιο το εργοστάσιο. Εγώ ήμουν στην ερευνητική ε, ομάδα για την περίπτωση ΑΖΕΝΤΕΦ ε, στην Γαλλία και σας έχω υποβάλει διάφορα σχόλια και ελπίζω να σας προσφέρω πολύτιμα στοιχεία κατά τη μελλοντική επεξεργασία της οδηγίας. Σε δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται διαρκώς οι μισθωτοί, ε, διότι όσο πιο ενημερωμένοι είναι, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουν για την αποφυγή ε, τέτοιων ατυχημάτων. Τέλος, πρέπει να αποφύγουμε τις ανθυπεργολαβίες, ε, γιατί τα μεγαλύτερα ατυχήματα σε αυτό οφείλονται στι μεγάλες βιομηχανίε σε μονάδες, ο εργολάβο, του υπεργολάβου, και τα κτλ. Οπότε ε, χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Εμείς είχαμε ζητήσει την απαγόρευση της ε, ε, διπλής και τριπλής υπεργολαβίας. Τέλο για την διαβούλευση, τη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να γίνει σαφής και σωστή αποτίμηση των κινδύνων και όχι να περιοριζόμαστε μόνο στον προσδιορισμό της περιμέτρου ασφαλείας αυτή η περίμετρο σε περίπτωση ατυχήματο και πυρκαγιά, κοιτάξτε, υπάρχει περίμετρο ασφαλεία που συνεπάγεται όμω ε, θύματα. Ε, χρειάζεται και περίμετρο μέσα ε, στο εργοστάσιο. Στην έρευνα που κάναμε όμω συνειδητοποιήσαμε ότι συχνά η περίμετρο ασφαλεία βρίσκεται μόνο εκτό του εργοστασίου για τους κατοίκους ε, της περιοχής ε, χρειάζεται ενημέρωση όταν υπάρχει κίνδυνος και για την εξωτερική περίμετρο αλλά και για την εσωτερική. Επίση, θα πρέπει να γίνονται προσωμιώσει ατυχημάτων για να ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να παραμείνουν ε, σε κλειστό χώρο, πρέπει να αποχωρήσουν. επίση ζώνες ε, ε, και ένωση και καταφύγια σε περίπτωση ατυχήματο και πυρκαγιά. Αυτά ανάντι θα πρέπει να προβλέπονται και να ρυθμίζονται. Για τη μεταφορά τώρα των επικίνδυνων ουσιών, όπω είπε και ο κ. Σένα, γίνονται μεταφορές... που ε- συνδέονται με αυτές τις ενδιάμεσες ζώνες αποθήκευσης όπως είπε ο εισηγητής. Αυτές μπορεί να είναι είτε μέσα στο εργοστάσιο είτε έξω από αυτό. Ε, στις, στους σταθμούς παραδείγματος χάρη βλέπουμε τρένα ολόκληρα που μεταφέρουν δεξαμενές ε, με έφλεκτα υλικά. Ε, ε, προφανέστατα τέτοια θέματα θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία. Ε, τρίτο πολύ σημαντικό θέμα η εποπτεία, ο έλεγχος. Ε, σε βέζο οδηγία λέτε. Ωραία. Εάν η οδηγία αν βάσει αυτή τη οδηγία θα πρέπει να γίνονται δύο επισκέψει το χρόνο τουλάχιστον. Ευνηδιαστική έλεγχη. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και αυτή οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι. Ένα τουλάχιστον. Εν τη αυτή περιπτώση, ο αριθμό των ελεγκτών, των επιθεωρητών, ε, θα πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού εγκαταστάσεων σε βέζο 3 τη χώρα αυτή. Ε, στη χώρα μου έχουμε πολύ λίγου επιθεωρητέ. Μα πώ να προλάβουν. Έχουν, υπάρχουν πάρα πολλέ εγκαταστάσει. Δεν έχουμε ε, αρκετό αριθμό επιθεωρητών. Η οδηγία λοιπόν, λοιπόν θα πρέπει να υποχρεώνει το κράτο μέλο, άρα κάνουμε συγκεκριμένη σύσταση εδώ, έτσι, να υποχρεώνει το κράτος μέλος ε, να αποφασίσει πόσου επιθεωρητές θα έχει σε συνάρτηση με τον αριθμό των εγκαταστάσεων που πρέπει να ελεγχθούν. Και ξαναλέω, δύο τουλάχιστον ευνηδιαστικέ επισκέψει σε όλε τι εγκαταστάσει στην επικράτεια τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Παναγιώτοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δύσκολη δουλειά της. Εγώ είμαι της και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή μας. Για την αναθεώρηση της οδηγίας σε Βέζο υπάρχουν τέσσερα κύρια σημεία τα οποία αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Επί τη ευκαιρία στο τελευταίο Στρασβούργο συζητήσαμε με τον κύριο Αντέρ, τον συγητή, τα ζητήματα αυτά. Η γενική μου άποψη είναι πως θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του περιβάλλοντος και των πολιτών χωρίς να ε, εμποδίσουμε την ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, σήμανση επικίνδυνων ουσιών. Η θέση μου είναι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ πέρα, η οποία βασίζεται σε ατυχήματα τα οποία έχουν ήδη συμβεί. Δεύτερον, λήψη αποφάσεων. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να επεκταθεί η συναπόφαση και στα παρατήματα 1 έως 7, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα της οδηγίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πράξη καταξιοδότηση τρίτων πληροφόρηση του κοινού. Υπάρχει η άποψη πως μπορεί μέσω της αντιπαράσεως διαδικτύου να αυξηθεί ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να ασχοληθούμε με, τα, με τους πραγματικούς κινδύνους, δηλαδή το ότι είναι πιο πιθανέ τα χημικά ατυχήματα από τρομοκρατική επίθεση και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι πληροφορημένοι οι πολιτέ μας. Τέταρτον, επιθεωρήσεις προτείνεται κάθε τρία χρόνια να υπάρχουν ε, μίνιμουμ κάθε τρία χρόνια έλεγχοι και μάξιμου ε, μάξιμουμ κάθε έτος. Συμφωνώ με αυτό, καθώς θεωρώ πως οι πόλεις οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες θα πρέπει να έχουν περισσότερους ελέγχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κομισιόν θέλει να πει δύο λογάκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε και δυνατότητα να πούμε λίγα λόγια σε σχέση με την πρόταση που υιοθέτησε η Επιτροπή και σε σχέση με τα σχόλια τα οποία έκαναν οι κύριοι και κυρίες βουλευτές. Πρώτα απ' όλα είναι ενδιαφέρον το ότι έχουμε εδώ πέρα μια αλλαγή η οποία ξεκίνησε από αλλαγή της κατάταξης των χημικών ουσιών. Ξεκίνησε αυτό από αναφορές σε ουσίες οι οποίες ε, υποβάλλονται στην ομοθεσία περί χημικών ουσιών και καθώς αλλάζουν οι κανόνες πρέπει, όπως λέει και η οδηγία, να προσαρμοστεί ο τρόπος αναφοράς ε, των ουσιών αυτών. Και βεβαίως ε, επί τη ευκαιρία η Κομισιόν κάνει μια πλήρη αναθεώρηση της οδηγίας. Το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν πως η οδηγία λειτουργεί καλά, έχει μειώσει τον αριθμό ατυχημάτων. Εάν δείτε την έκθεση εφαρμογής που δημοσιεύτηκε θα δείτε πως παρά την αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων που έχουν καταγραφεί στην Ένωση, ο αριθμός σοβαρών ατυχημάτων μειώνεται. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πως υπάρχουν αρκετά ατυχήματα. Είναι πολύ υψηλός αυτός ο αριθμός και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το μέσο αυτό σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να αποφύγουμε αυτά τα ατυχήματα και να περιορίσουμε τις συνεπίες τους. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην ε, κατάταξη των χημικών ουσιών και το γιατί προτείναμε μια εργαλειοθήκη για να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από κάποια ευελιξία. Είναι οι κανόνες ε, περί χημικών ουσιών σημαίνουν πως κάποιες χημικές ουσίες ε, στο μέλλον θα κατατάσσονται με βάση τις ε, εγγενείς τους ιδιότητες και άρα θα υπάγονται στην οδηγία σε βέζο. Η πείρα μας δείχνει πως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες οι εγγενείς αυτές ιδιότητες μιας ουσίας δεν αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στις συνθήκες χρήσης αυτών των ουσιών από τη βιομηχανία. Και για τις περιπτώσεις αυτές η Κομισιόν έχει προτείνει την δυνατότητα υιοθέτηση πράξεων κάτω εξουσιοδότηση που θα ορίζουν ε, τους όρους ε, κατά τους οποίους θα καλύπτονται αυτές οι ουσίες από την οδηγία ε, έτσι ώστε να επικεντρωνόμαστε στο όταν εμφανίζονται κίνδυνοι. Και θεωρούμε πως το κατάλληλο μέσο γι' αυτό είναι πράξεις κατεξιοδότηση. Να επισημάνω πως η κατάταξη των χημικών ουσιών σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας σύμφωνα με τα ορίζει η συνθήκη. Οπότε θεωρούμε πως δευτερογενής νομοθεσία εδώ πέρα είναι ο κατάλληλος τρόπος για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε λεπτομερώς περιπτώσεις στις οποίες αυτές είναι ο καταταγής ουσίες θα επηρεάσουν το πεδίο εφαρμογή σε ΣΕΒΕΖΟ. Να πω εδώ πέρα πω δεν μιλάμε για μια γενική προσέγγιση, θα είναι μια προσέγγιση κατά εξαίρεση με βάση κριτήρια που θα οριστούν στο παράρτημα 7 τη οδηγία. Θεωρούμε πω αυτό είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της οδηγίας που εξασφαλίζει αναλογικότητα των ε, παρεμβάσεων των ρυθμιστικών και τον αντίκτυπο στη βιομηχανία και ε, τη μεγαλύτερη ασφάλεια του κοινού. Όσον αφορά το θέμα των φυσικών καταστροφών που ανέφερε ο εισηγητής. Το παράδειγμα 2 ορίζει το τι πρέπει να περιέχει το βασικό μέσο. Και αυτό έχει εισαχθεί σε αυτή την οδηγία, αλλά τα σενάρια τα οποία εξετάζουμε πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες και σεισμούς. Οπότε έχουμε συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο, το οποίο συμφωνούμε μαζί σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, ε, έχουμε εισαγάγει ένα συγκεκριμένο σημείο για την εξέταση παλαιών ατυχημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Και μάλιστα το θέμα αυτό, η εξαγωγή συμπερασμάτων, είναι κάτι το οποίο έχουμε ενισχύσει ιδιαίτερα, όχι μόνο εδώ πέρα, αλλά και μέσω των κρατών μελών που είχαν σοβαρά ατυχήματα για να μοιράσουν ε, αυτή τη γνώση τους. Βλέπω πως θέλετε να τελειώνω, να αναφερθώ σε κάποια άλλα σημεία, αν μου επιτρέπετε, που είπε ο εισηγητής. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Να πω πως όσον αφορά την ανάμειξη των εργαζομένων, υπήρχε μια τροπολογία μετά το ατύχημα της Τουλούζης και η τροπολογία αυτή εισήγαγε την εμπλοκή των εργαζομένων στο σύστημα διαχείρισης ασφαλείας και την εμπλοκή των εργαζομένων στα εσωτερικά σχέδια άγγης. Όσον αφορά τις μεταφορές, οι μεταφορές ρυθμίζονται από ειδική νομοθεσία που ενισχύθηκε το 2008 και αναφέρεται σε οδικές, συντηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Θεωρούν πως είναι διαφορετικοί κανόνες που πρέπει να ισχύσουν για τις μεταφορές γιατί τα μέσα του ΣΕΒΕΖΟ αφορούν ειδικά σταθερές εγκαταστάσεις. Δεν είναι ο ίδιος κίνδυνος λοιπόν που αντιμετωπίζουμε, ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλότερος και να απαιτεί πιο συγκεκριμένη νομοθεσία. Νομίζω πως απάντησα κύριε Πρόεδρε σε κάποια σημαντικά ερωτήματα, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τον λόγο στους ε, σκιοδησηγητές αν θέλετε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το κλίμα που επικρατεί, που διαπιστώνω από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και βλέπω μια σχετική ομοθυμία δεν συμφωνούμε απολύτως με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό είναι ο ρόλο μας, να προσπαθούμε να επηρεάζουμε τις εξελίξεις. Ε, δεν θέλουμε βεβαίω να περιορίσουμε την βιομηχανία. Πρέπει να παράγει αυτά που χρειάζεται η κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κατοχυρώσουμε την ε, ασφάλεια των ε, συμπολιτών, του περιβάλλοντος, τη κοινωνία. Ήσασταν πολύ σύντομο. Σα ευχαριστώ το χρονοδιάγραμμα το έχετε. Περνάμε στο επόμενο σημείο, 7. Μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση ομαδικών πρόσφυγων. Η κυρία Κολάρσκα Βομπίνσκα είναι η συγγήτρια και έχει άρα το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συζήτηση για τις συλλογικέ αγωγές, ε, τις συλλογικέ επανορθώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καινούρια για μας το 2008 λάβαμε την πρώτη λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις συλλογικέ επανορθώσεις για τα antitrust τη δράση αντιτράστα και επίσης για τις συλλογικές προσφυγές των καταναλωτών. Το 2009 το Μάρτιο υιοθέτησε το Κοινοβούλιο ένα σχετικό ψήφισμα και τώρα μόνο και δυνάμει της συνθήκη της Λισαβόνας Επανερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προχωρήσει προς την υιοθέτηση νομοθεσίας και άρα ξεκίνησε την διαβούλευση και θα συμμετάσχουμε και εμείς στη διαβούλευση. Η έκθεση αυτή νομίζω θα επιβεβαιώσει την προηγούμενη θέση του Κοινοβουλίου και θα σε εξηγήσω γιατί. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αποσαφηνίσω τη βασική μου θέση γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό και πιστεύω ότι θα προκύψει και μια διάσταση απόψε, μια διχογνωμία. Πρέπει να αναρωτηθούμε για δύο πράγματα. Πρώτον, επιθυμούμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, συλλογική επανόρθωση. Ε, γνωρίζουμε ότι λειτουργεί ένα σύστημα, ένα αντίστοιχο σύστημα στι ΗΠΑ και πρέπει να αναρωτηθούμε, θέλουμε ένα παρεμφερέ σύστημα στην Ευρώπη. Δεύτερον, εάν ναι, τι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει, ποιοι πρέπει να είναι οι περιορισμοί του συστήματος αυτού. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ναι, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα και καλωσορίζω τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, θεσμοθετήσει ε, αποτελεσματικά ένδικα μέτρα για όλους όσους παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Ε, όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε για τους περιορισμούς ως προς τους καταναλωτές και ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να προστατευθούν Ποιο είναι το θέμα. Οποιοδήποτε σύστημα είναι να, πρέπει να λειτουργεί και για τις μικρές επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές και όχι να δίνει άλλο ένα μέσο στις μεγάλες εταιρείες για να αλληλομηνύονται ε, γιατί ορισμένες φορές δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα λόγω αυτού Εννοεί ότι χρειαζόμαστε ισχυρές δικλείδες ε, ασφαλείας ε, για να προστατεύσουμε κάποιες επιχειρήσεις κατά της καταχρηστικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών. σε, για τις αγωγέ αυτές. Δεν θέλουμε ξαφνικά να προκύψουν επαγγελματικέ οργανώσει που θα καταθέτουν αυτές τις συλλογικέ αγωγέ. Δεν επιθυμούμε να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα που θα δημιουργήσει κέρδη και μόνο και μόνο γι' αυτό να γίνονται ε, οι αγωγέ. Δεύτερον, θα πρέπει να εγγυηθεί ότι θα καλύπτει διαστική ευθύνη για τις δαπάνες ε, της δίκης. Ε, τρίτον, οποιαδήποτε αγωγή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης για το παραδεικτό πριν ε, αρχίσει η δημόσια ακρόαση. Τέλος, χρειαζόμαστε τους κανόνες για τη δικαιοδοσία. Να αποφύγουμε το υπονομαζόμενο forum shopping, δηλαδή την επιδίωξη του ευνοϊκότερου εφαρμοστέου δικαίου ε, για να μην ε, ή με για να μην στρέφεται ο ε, ενάγων προς μια άλλη χώρα που ναι δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της δίκης αλλά έχει ευνοϊκότερο εφαρμοστέο δίκαιο. Άρα χρειαζόμαστε σαφέστερη διατύπωση για, τις, ε, για το θέμα αυτό. Υποστηρίζω την προηγούμενη θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή η αδίποτε συμμετοχή σε ε, συλλογική αγωγή θα πρέπει να υπόκειται σε αίρεση opt-in για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίση θα πρέπει να είναι αναλογικό το σύστημα ώστε τα κράτη-μέλη, τα μονομένα κράτη-μέλη να έχουν περιθώριο ελιγμών για να προσαρμόσουν την ε, κείμενη νομοθεσία του ε, ε, οποιαδήποτε. Τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε ελάχιστα πρότυπα και σε θελοντικέ κατευθυντήριε γραμμέ για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα ένομα συστήματα των κρατών μελών κατόπιν θα εφαρμόσουν τι διατάξεις αυτό θα καλύπτει και τις αποζημιώσεις Φυσικά αυτό το θέμα είναι λεπτό διότι ε, πρόκειται για οικονομικό ζήτημα και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι εθνική αρμοδιότητα ε, το θέμα της αποζημίωσης. Ε, τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε επαρκή νομική βάση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τις συλλογικέ επανορθώσεις και θα πρέπει ε, να γνωμοδοτήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα που προανέφερα πριν ναι, προχωρήσουμε. Τέλος, ο βασικός στόχος του συστήματος θα πρέπει να είναι να διευκολύνει την ε, πρόσβαση, την προσφυγή στη δικαιοσύνη και για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σαφές όμως από την εμπειρία που έχουμε σε χώρες που ήδη λειτουργεί τέτοιο σύστημα ότι οι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών είναι ταχύτεροι και συνεπάγονται χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την υποβολή αγωγής. Καλούμεθα λοιπόν να επιλέξουμε το δρόμο που θα ακολουθήσουμε και να θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και το εξή. Ο εναλλακτικό μηχανισμό ε, επίλυση διαφορών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να ε, έρονται οι διατάξει όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίζουν πώ θα κινηθούν. Υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπω σα έλεγα στην αρχή και εύχομαι στην Επιτροπή μας να κάνουμε μια εισβάθος συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Όχι, De Angelis. Ε, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μορφές συλλογικής προσφυγής που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη είναι αρκετές και πολλές φορές υπάρχουν και αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Δεν υπάρχει κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν δύο συστήματα τα οποία να είναι ε, ταυτόσημα στα κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλήττονται οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούν να υποφεληθούν από ένα σύστημα κοινό και υπάρχει αβεβαιότητα και για τι επιχειρήσει. και υπάρχει και κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα αυτό. Το 2005 και το 2008 εκδόθηκε μία πρώτη λευκή βίβλος, ε, ε, η πράσινη βίβλο και οι θέσεις που εκφράζονται είναι σαφείς για τους ε, καταναλωτές, δεν ε, συμφωνούσαν όμως οι επιχειρήσεις. Είναι θέματα αρκετά ευαίσθητα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη νομική παράδοση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθήσουμε ήδη υφιστάμενες διαδικασίες για θέματα προσφυγής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών, όπως είπαμε, και αυτή η διαδικασία μπορεί να ισχύσει σε μεμονωμένους μονοτομεί σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά κράτη-μέλη ε, αφήνουν ε, ε, στις εθνικέ αρχές τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγέ, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη μπορούν οι οργανώσεις καταναλωτών να αναλάβουν δράση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες όσον αφορά τα θύματα περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να ισχύσει συλλογική προσφυγή. Μια πολύ διαφορετική λοιπόν κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη, κάτι το οποίο θίγει και αυτά τα οποία περιμένουμε από μια εσωτερική αγορά. Όπως βλέπετε και από το χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλουμε να διευκολύνουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, να έχουν ε, κοινή αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη, αλλά δεν ξέρω αν ε, ένα κοινό τρόπο συλλογική προσφυγή είναι το κατάλληλο μέσο. σω να υπάρχει κάποια άλλη μέθοδο που να είναι και πιο γρήγορη και πιο φθηνή όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όμω το θέμα τη συλλογική προσφυγή είναι θέμα για το οποίο έχουν δοθεί ιστορικέ μάχε για τα δικαιώματα των καταναλωτών και ίσω έχει φτάσει η στιγμή για να βρεθεί μια εγγύηση για τα δικαιώματα δικαιώματα των καταναλωτών και να είναι και κάτι που θα θεωρείται από όλους τους εμπλεκομένους μια λογική λύση. Είναι απαραίτητο να βρεθεί μια λύση στην οποία θα συμφωνούν και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις των καταναλωτών ε, και οι μικροεπιχειρήσεις. από την ομάδα μας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, επιφυλάσσομαι προς το παρόν για να στείλουμε τις ε, παρατηρήσεις μας προς τον εισηγητή ούτως ώστε να μπορέσει προς την εισηγητή συγγνώμη, ούτως ώστε να έχουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σαφώς χρειάζεται να επιτευχθεί μια πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, την, για το θέμα της συλλογική προσφυγής και χαιρετίζω τα σχόλια της εισηγήτριας, ιδίως όσον αφορά ε, τα σημεία στα οποία θα υποφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη βρίσκονται σε δύσκολη θέση όταν θα πρέπει ε, να υποβάλουν χωριστές αγωγές. Ε, είναι αδύναμη η θέση τους έναντι των μεγάλων πολυεθνικών. Και νομίζω ότι ω τμήμα των προσπαθειών μα να υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα πρέπει να εξετάσουμε θετικά τη δυνατότητα η οποία προσφέρεται να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να συνεργάζονται στο πλαίσιο μια συλλογική προσφυγή. Και για του καταναλωτέ εξάλλου, υπάρχει μια δυνατότητα, ιδίως ε, στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου, διότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές στι διάφορες χώρε να ασκήσουν μια κοινή αγωγή και αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν αγοράζουν κάτι από το διαδίκτυο παραδείγματο χάρη ή αν πληρώσουν για παροχή κάποιας υπηρεσία στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ να, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνενώσουν τις προσπάθειές τους ε, σε μια κοινή δράση με τη συλλογική προσφυγή θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά, κάτι το οποίο θα είναι προς όφελος των εταιριών που θέλουν να αναπτυχθούν σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να προσθέσω ακόμη σε αυτά τα οποία είπε η συγγήτρια ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν για περιβαλλοντικές δράσεις ε, είναι σημαντικές. Υπήρξαν αρκετά περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπήρξε κάποιο ατύχημα, υπήρξε κάποιο ε, περίπτωση ρήπανσης, όπου δεν πλήττεται μόνο ένα κράτος μέλος, πολλές περιφέρειες από διαφορετικά κράτη-μέλη μπορεί να πλήττονται από ατυχήματα και πρόσφατα είχαμε ε, το παράδειγμα ε, της ε, Ερυθράς ηλίου στην Ουγγαρία που επηρέασε το Δούναβι και όλες τις χώρες από τις οποίες περνούσε ο Δούναβης και είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορέσει να αναλυθεί δράση σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία αγορά, γιατί εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, σκοπός ε, μας είναι να δημιουργηθεί ένα δίκαιο πεδίο στο οποίο να μπορούν να επωφελούνται ε, ή να επιβαρύνονται από το άχθος όλοι εξίσου και αν συμβεί κάτι είναι δύσκολο να έχουμε μέτρα επανόρθωσης, πράγμα το οποίο θέτει φραγμούς για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και δεν μιλάω μόνο για την αποζημίωση, αλλά και για ασφαλιστικά μέτρα που θα πρέπει να μπορούν να ληφθούν, ώστε ε, να σταματά μια συγκεκριμένη δράση μια εταιρεία, παραδείγματο χάρη, που θα είναι ει βάρο των καταναλωτών των επιχειρήσεων. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και για την προστασία του περιβάλλοντος και για να έχουμε μια νέα αγορά και για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στις δύσκολες λεπτομέρειες και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κύριος Τούρμες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση εδώ πέρα γιατί είναι και καυτό πολιτικό θέμα. Όσοι είναι καιρό στο Κοινοβούλιο θα θυμούνται πως υπήρχε μια αρχική πρόταση της Κομισιόν το 2005 που ήθελε να δώσει τέτοιες δυνατότητες ομαδικών πρόσφυγων, ειδικά σε περιπτώσεις πολυεθνικών εταιριών, η οποία τότε δεν πέρασε. Ε, υπό την ηγεσία του κυρίου Λένε, που και πάλι τώρα κατά βάση είναι ο εισηγητής στην κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή. Ως πράσινοι θεωρούμε πως πρέπει να βρεθεί ένα συμβασμός ώστε αφενός να μην πάμε σε κάποιες από τις καταχρήσεις που έχουμε στη ΣΥΠΑ γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε ε, κυρίως οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με μαζικές τέτοιες προσφυγές μπορούν να κερδίσουν τεράστια ποσά και συχνά πολύ περισσότερα από τους καταναλωτές στο τέλος από τους οποίους υποτίθεται πως ε, εκπροσωπούν. Χρειάζεται μία λύση γι' αυτό. Δεν έχω λύση, αλλά την ψάχνουμε. Δεύτερον, συμφωνούμε με τους φιλελεύθερους και την κυρία Χολ πως ε, πρέπει να διευκολυνθούν ομαδικές προσφυγές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και βεβαίως αυτό θα ισχύει για τους καταναλωτές στην Ευρώπη και τις αγορές οι οποίες ε, ε, πλέον ενοποιούνται ειδικά αγορά ηλεκτρονικών κτλ. Οπότε χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στον τομέα αυτόν. Κατά βάση αυτά. Και αναμένω βεβαίω στη συνεργασία με την κυρία Μπομπίνσκα. Αγγέλικα Νίμπλερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εισαγωγή. Εδώ και χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι πάρα πολύ εντατικά βεβαίω, αλλά συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τούρμες πως εγώ αυτό το θέμα το συνδέω πρώτα απ' όλα με το σύστημα που υπάρχει στη ΣΥΠΑ και ως δικηγόρος ε, τρομάζομαι αυτά τα πράγματα γιατί στη ΣΥΠΑ πραγματικά αυτά αποτελούν μια τεράστια μηχανή παραγωγής χρήματος για τους δικηγόρους που ασχολούνται με αυτά. Αλλά δεν έχει στόχο αυτό τον οποίο θέλουμε εμείς, δηλαδή με τις ομαδικές ε, προσφυγές δεν ε, ενισχύεται το σύστημα προστασίας του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε τι περιορισμούς ε, θα εισαγωγούμε εδώ πέρα για να μην υπάρχουν καταχρήσεις ε, του συστήματος. Ξέρετε τις συνέπειες ε, λόγω των πληρωμών ύψους εκατομμυρίων που πηγαίνουν σε αυτούς που κάνουν τις αγωγές και στους δικηγόρους τους και το αποτέλεσμα ήταν ένα σε όλες τις ε, πληροφορίες, σε όλες τις εγγυήσεις προϊόντων, στις πληροφορίες στον καταναλωτή. Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσει οι οποίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Ε, δηλαδή μη βάλετε το κεφάλι σας στο πλυντήριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι προφανές. Αλλά επειδή κάποιος πήγε και έκανε μια αγωγή, υπάρχει τώρα μια τέτοια προειδοποίηση. Σαν πλυντήρια, ξέρω εγώ, στις είπα. Οπότε δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιες καταχρήσεις και βεβαίως ε, χαίρομαι για το ότι προσεγγίζει κάπως διαφορετικά το θέμα η συγκήτρια, αναγνωρίζει πως υπάρχουν κάποιες αναγκαιότητες εδώ πέρα και υπάρχει βεβαίως, ε, θα πρέπει να διηγηθούμε σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, αλλά να λάβει υπόψη παρακαλώ και την δική μας ε, γνωμοδότηση της δικής μας επιτροπής πως υπάρχουν φοβερές δυνατότητες κατάχρησης. Δεν είναι θεωρητικά αυτά. Δείτε την ομολογία στη ΣΥΠΑ. Δεν θα πρέπει να προσαρμόσουμε το σύστημά μας σε αυτό τον, τον ΙΠΑ. Αλλά δεν νομίζω πως αυτό θέλουμε ε, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γκέμπελς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσωπικά, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι κατά ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, συλλογικών, ε, συλλογικής προσφυγής. Άκουσα μέσω, με μεγάλη προσοχή τους συναδέλφους ε, που επιθυμούν να υπερασπιστούν το περιβάλλον, ε, να ταχθούν κατά των πολυεθνικών, ε, να υπεραμεινθούν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, των ορφανών και χειρών, αλλά ωραία όλα αυτά. Η πραγματικότητα όμως είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ας δούμε τι γίνεται στις ΙΠΑ, από που προέρχεται το σύστημα. η μεγάλη, τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία ψαρεύουν ενάγοντες και στην πλάτη τους κερδοφορούν όταν κερδίζουν τη δίκη. Τέτοιο σύστημα εγώ προσωπικά δεν θέλω να θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορέσετε να το αποφύγετε αν επιτρέψετε την ε, συλλογική προσφυγή. Πώς λέει θα το κάνετε, θα πείτε ότι πώς θα αποδείξετε ότι είναι προς συμφέρον των καταναλωτών της κοινωνίας ή δεν ξέρω εγώ νου άλλου αν επιτρέψετε ένα τέτοιο σύστημα συλλογικής αγωγής ή έχουμε ή δεν έχουμε σύστημα. Αν υπάρχει θα υπάρξουν και καταχρήσεις εγώ προσωπικά πιστεύω πως δεν πρέπει να εισαγάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλους παραλογισμούς και τα λάθη του Αμερικανικού συστήματος δικαιοσύνης. Ας τα αφήσουμε στην επικουρικότητα. Αν θέλουν κάποιοι που θέλουν να το οργανώσουν, ας το οργανώσουν. Υπάρχουν κάποιοι εδώ, φίλος μου πίσω, που το έχουν ήδη κάνει. Γιατί να μην είναι θέμα επικουρικότητας. Δεν κρίνω ότι χρειάζεται ρύθμιση σε επίπεδο ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαίρω την Επιτροπή που δρομολόγησε τη διαβούλευση διότι πραγματικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ζήτημα και είναι ένα ουσιαστικό ε, πολιτικό πρόβλημα. Ή θα τους αφήσουμε στη μοίρα τους τους πολίτες, ε, μπορούμε να μιλήσουμε για τους καταναλωτές αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις, μπορούμε λοιπόν να τους αφήσουμε όλους αυτούς απροστάτευτους ενώπιον των πολυεθνικών που έχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα στη διάθεσή τους Μόνοι μόνος του κανείς δεν μπορεί τίποτα να κάνει κατά τις πολυεθνίκες. Θα σας δώσω εγώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι μεγάλες ε, φαρμακευτικές εταιρείε. Αν σας πουλήσουν ένα φάρμακο που έχει σοβαρές παρενέργειες, με ποιο τρόπο εσείς, ο μικρός πολίτης, που έχετε αρρωστήσει ε, χρησιμοποιώντας το φάρμακο θα επιτεθείτε κατά της ε, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν γίνεται αυτό. Ε, λοιπόν, τώρα για το σύστημα το αμερικανικό, για τις class actions, τις συλλογικέ αγωγές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η Apple έβγαλε το iPad, το iPad δεν είχε μπαταρία, δεν μπορούσε κανεί να την αντικαταστήσει. Έγινε λοιπόν η συλλογική αγωγή, νίκησαν και δύο χρόνια μετά η νέα εκδοχή του iPad ε, είχε μπαταρία ε, που μπορούσε κανείς να αλλάξει, να αντικαταστήσει. Βλέπετε λοιπόν ε, πόσο ο καταναλωτής ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη εταιρεία και με ένα σπάρο δύο τριγώνια. συγγνώμη, αλλά, κα, την, την ΣΥΠΑ, αλλά ή μάλλον να στο πω αλλιώς για το σύστημα συλλογική αγωγή, ε, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα ε, δικό μας ευρωπαϊκό σύστημα να ομαδοποιούνται οι καταναλωτέ. οι μικρόμεσες επιχειρήσεις και σε επίπεδο δικηγορικού ε, γραφείου θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο για να μην παίρνουν υπέρογγε αμοιβέ όταν κερδίζουν τη δίκη αλλά ε, ήδη υπάρχει μια τέτοια διαδικασία σε διάφορα ένομα συστήματα, ενώ εμείς στην Ευρώπη δεν τονώνουμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τη δράση που μπορούν να αναλάβουν κατά των πολυεθνικών εταιριών. Donc, je pense que utile, Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αντίστοιχο θεσμό στην Ευρώπη και ενθαρρύνω τον εισηγητή να ε, προτείνει ε, την υποστήριξη αυτής της οδηγίας διότι προστατεύει τον καταναλωτή και τις μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Μήπω ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει σύντομα το λόγο. Ένα-δύο λεπτάκια έχουμε και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω ε, Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαρκή ε, συμμετοχή στο διάλογο και στη διαβούλευση που έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. Τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Κοινοβουλίου. Τώρα επιδιώκουμε να βρούμε κοινέ αρχές για τις ε, συλλογικές αγωγές σε οποιοδήποτε πεδίο της νομοθεσίας της Ένωσης. Κοινέ αρχές λοιπόν για συλλογικές αγωγές για να διακοπεί η παράνομη παράνομη, να τερματιστεί η παράνομη συμπεριφορά ή ε, σε περίπτωση παραβίαση νομοθεσία ε, για τη διεκδίκηση αποζημίωση. Και ιδιαίτερα το δεύτερο κομμάτι, αυτό το δεύτερο κομμάτι τη διαβούλευση οδηγεί σε εντονότατε συζητήσει, διότι αυτόματα όλοι σκέφτονται το σύστημα class action, δηλαδή συλλογική αγωγή των ΗΠΑ. Σα διαβεβαιώ ότι αυτό είναι το τελευταίο που θα θέλαμε να θεσπίζετε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε αντίστοιχη κουλτούρα ω προ τη διευθέτηση των διαφορών, όπω δηλαδή στη ΣΥΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει δεν υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσει. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα και αυτό επιζητούμε σήμερα. Να επιτύχουμε τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα αφενό ε, στην δυνατότητα των θυμάτων μετά από παραβίαση τη νομοθεσία τη Ένωση και πρόκειται για ιδιώτε ή μικρομεσαίε επιχειρήσει, να του επιτρέψουμε λοιπόν να διεκδικήσουν την αποζημίωση που δικαιούνται και αφετέρου να μην πέσουμε στην παγίδα του συστήματος των ΗΠΑ όπου έχουμε κατάχρηση ουσιαστικά του συστήματος, καταχρηστικές αγωγές. Ε, πρέπει να βρούμε λοιπόν δικλείδες ασφαλείας και μπορούμε να εμπνευστούμε από τα υφιστάμενα εθνικά ένομα συστήματα και χαιρόμαστε που σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα διερευνήσουμε τις εναλλακτικέ ε, λύσεις που έχουμε. Να σας πω ότι δύο εβδομάδες μετά το πέρας της δημόσιας ε, διαβούλευσης σήμερα δεν μπορώ να κάνω μια επισκόπηση ε, των αποτελεσμάτων διότι λάβαμε σχεδόν 300 απαντήσεις, δηλαδή 4.000 σελίδες από ενώσεις επιχειρήσεων, καταναλωτών και δικηγορικά γραφεία κυρίως. Και 18.000 πολίτες πέραν αυτού επίσης μας έστειλαν επιστολή. Ε, ευελπιστούμε λοιπόν στο εγγύ μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στην Επιτροπή σα και να σα ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα τη διαβούλευση. Στο μεταξύ αν υπάρχουν ερωτήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ στη διάθεσή σα. είμαι. Ευχαριστώ πολύ και την άλλη μια φορά το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Sorry. As you have seen, even right now... Όπως είδατε, ακόμη και τώρα, κάποια μέλη της Επιτροπής μας λένε ότι δεν χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα συλλογικής προσφυγή, ενώ άλλοι συνάδελφοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε. Βλέπετε ότι υπάρχουν λοιπόν πραγματικά ουσιαστικές διαφορές. Πριν περάσω σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουμε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Και θα πρέπει να συνοψιστεί όλη η συζήτηση που θα έχει γίνει με τη δημόσια διαβούλευση και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα γιατί είναι ένα θέμα δύσκολο και πολύ πολιτικό. Αν συμφωνείτε λοιπόν αυτή είναι η σωστή άποψη κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου ένα ευρωπαϊκό σύστημα είναι απαραίτητο. Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και με την κοινή ευρωπαϊκή αγορά χρειαζόμαστε και ε, δυνατότητα για τον καταναλωτή να μπορεί να υπερασπίζεται τη θέση του, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το σύστημα προσφυγών δεν είναι κάτι το οποίο εμποδίζει την ενιαία αγορά, αλλά είναι ένα γενές τμήμα της αγοράς. είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τις επιχειρήσεις ε, με στόχο την ανάπτυξη της κοινή αγοράς. Σε ένα σύστημα στο οποίο όλοι θα επωφεληθούν όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ διαφορετικά τα νομικά συστήματα στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν χώρες, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν κανένα θεσμικό όργανο που να ασχολείται με συλλογικές προσφυγές. Παραδείγματος χάρη η Πολωνία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να οργανώσει ένα εντελώς νέο σύστημα για να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Και θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση σε αυτό τον τομέα του δικαίου γιατί θα πρέπει τα διοικητικά δικαστήρια να λάβουν νέες τέτοιε αποφάσεις. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα. Τώρα κάποιε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Η κυρία Χόλ ανέφερε κάτι το οποίο θα επανέλθει στις συζητήσεις μας, το θέμα των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παραδείγματο χάρη ε, το, το θέμα της ρήπανσης στο Δούναβι. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάποια στιγμή πώς το βλέπετε εσείς. Οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών θα αναλάβουν συλλογική δράση κατά μία εταιρεία που δημιούργησε μια οικολογική καταστροφή σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, ένα νέος προβληματισμός και αν αρχίσουμε τέτοιου είδους συζητήσεις δεν θα βρούμε τελικά συμφωνία σε πολύ βασικά ζητήματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Το βλέπω και εγώ το πρόβλημα αυτό που αναφέρατε. Ε, τι θα γίνει σε περίπτωση μιας καταστροφής ε, όπως της ε, Φουκουσίμα που μπορεί να συμβεί στα σύνορα μιας χώρας και να επηρεάσει πάρα πολλές χώρες. Ποιος θα ασκήσει προσφυγή εναντίον τίνος για να καλυφθεί το κόστος. Θέλω να πω ότι αν ξεκινήσουμε τέτοιου είδους συζήτηση, δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία για κάποια βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Είναι μια εντελώ νέα κατάσταση, νέα προβλήματα και θα ήθελα να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία ήδη θεωρούμε σημαντικά. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σα και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα τη δημόσια συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία συνάδελφε. Τελειώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχουμε και λίγο χρόνο ε, είχαμε λίγο χρόνο για τι συζητήσει και άρα ξεκινήσει η συζήτηση. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερικής διάταξη το υπαριθμό 8 και... ορίζω την κυρία Χέντεγκαρντ και βεβαίως θα ακούσουμε από εκείνη πρώτα απ' όλα πώς πάνε οι υποθέσεις της και δε βεβαίως μετά θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις, να πούμε και τίποτα και εμείς κάνουμε κάποιες υποδείξεις και έχουμε προβλέψει χρόνο για να έχουμε κάποια βάση για τη συζήτησή μας. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ευχαρίστηση να έρχομαι στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, και Έρευνας και Ενέργειας στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Στους πρώτους πέντε μήνες του έτους η Κομισιόν ε, συνέχισε να θέτει τα θεμέλια του πιο φιλόδοξου προγράμματος στον κόσμο για την κλιματική αλλαγή και προβλέπουμε και άλλη δράση ε, φέτος. Όπως ξέρετε η κλιματική αλλαγή αφορά και την ενέργεια, την ενεργειακή ασφάλεια και το πώς θα έχουμε πολιτικές οι οποίες θα αποτελέσουν κίνητρο για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας πρώτα απ' όλα για τον οδικό χάρτη του 2050 και το πώς θα πάμε πέρα από το 20%. Όπως ξέρετε το Μάρτιο υιοθετήσαμε το οδικό χάρτη του 2050 για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος προετοιμάζει προτάσεις για υιοθέτηση στις 21 Ιουνίου και αναμένουμε βεβαίως πρωτοβουλίες ε, του Κοινοβουλίου. Αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο των πρωτοβουλειών για το 2020 και υποστηρίζει τους ε, στόχους ενέργειας και κλίματος και πάει πέρα ε, από τον ορίζοντα του 2020 για το πώς μπορεί η Ένωση να πετύχει τους στόχους της και να μειώσει τις εκπομπές μέχρι 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα σε σύγκριση με το 1990 και να δούμε και τι κάνουν γενικά οι ανεπτυγμένες χώρες. Καλώς ορίζω το έργο που κάνει η Επιτροπή σας στην γνωμοδότησή της που υιοθέτησε πρόσφατα επίσης ε, αναφέρει συστάσεις που υπήρχαν ε, στην ανάλυση των επιλογών για να πάμε πέρα από το 20% και να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Ξέρουμε πως μεταξύ των πρακτικών μέτρων που θα μπορούσε να αναλάβει η Κομισιόν συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη επαρκών πόρων για το σχέδιο αυτό και χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως τα σχέδια τα οποία θα τρέχουν συνεχώς. Οπότε εξετάζουμε τις προοπτικές του 2050 και κοιτάμε πώς θα κινητοποιήσουμε πόρους σήμερα για να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και φιλική στον άνθρακα σήμερα και μακροπρόθεσμα. Οπότε αναμένω βεβαίως ε, και τις αποφάσεις ολομέλειας του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Να αναφέρω κάτι για το 2050 τον οδικό χάρτη. Δύο σημαντικά πράγματα πρέπει να ξέρουμε. να είναι πως εισάγουμε εδώ πέρα μια αλλαγή προτύπων αυτό το οποίο κάνουμε μέχρι στιγμή στην Ευρώπη είναι να κάνουμε δεσμεύσεις μέσω αντιστάθμισης. Αγοράζουμε δηλαδή πράγματα κυρίως στην Κίνα, Ινδία, Κορία, Κορέα, Ινδονησία και Βραζιλία. Με άλλα λόγια, δίνουμε λεφτά στους ανταγωνιστές μας. Αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει ως μακροπρόθεσμη στρατηγική πώς είναι καλύτερο να επενδύσουμε στην ίδια την Ευρώπη και στη δική μας καινοτομία αντί για τους ανταγωνιστές. Και επίσης λέει ε, σαφώς πως δεν θα μπορέσουμε πλέον να αγοράσουμε τίποτα άλλο σε άλλες περιοχές γιατί τα φτηνά θα τα κάνουν μόνοι τους, δεν θα τα δώσουν ε, σε ευρωπαϊκές χώρες οι εταιρείε. Αυτό είναι το, το άλλο στοιχείο μετά ε, όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτήν, στον οδικό αυτό χάρτη και μπορούμε να αποδείξουμε πως ε, αρκεί η Ευρώπη να έπαιρνε στα σοβαρά αυτό το στόχο του 20% αυτό από μόνο του θα μας πήγαινε πέρα από τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 20% και γι' αυτό λέμε πως για να ασχοληθούμε ειδικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα ειδικά στον τομέα των κτηρίων που μπορεί να δημιουργήσει και δουλειές ε, στον τομέα των κατασκευών που έχει υψηλή ανεργία θα ε, μας εξυπηρετήσει κιόλας. Θα δημιουργήσει δουλειές που δεν μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό, π.χ. στην ανακαίνιση κτηρίων. Να πω λίγα λόγια για την περαιτέρω εφαρμογή του πακέτου κλίματος και ενέργειας. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι βεβαίως η ναυαρχίδα μας εδώ πέρα θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση του 2013. Όλα τα απαραίτητα μέτρα προετοιμάζονται για να υπάρξει μια ήπια μετάβαση και αυτή τη στιγμή βεβαίω ε, ετοιμάζονται τα εφαρμοστικά μέτρα. Πιο τεχνικά τέτοια μέτρα επίσης προβλέπονται για να υιοθετηθούν πριν το τέλος του 2011 μετά τα πρόσφατα γεγονότα που θα έχετε παρατηρήσει με τα αρχεία του συστήματος εμπορίας εκπομπών υπάρχει τεράστια προσπάθεια από τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να, υπάρξει, να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας χωρίς τις οποίες δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν τα μητρώα τους οπότε εξετάζουμε αυτά τα μέτρα και μαζί με τους ενδιαφερομένους εξετάζουμε και μέσο πρόθεσμα της ε, πρωτοβουλίες και θα ξέρετε πως μετά θα έχουμε μια πιο ενιαία πλατφόρμα ε, για να γίνονται οι δημοπρασίες. Βεβαίως μετά έχουμε ως σημείο κλειδί το πολιετές πλαίσιο το οποίο Μα απασχολεί. Θα παρουσιάσουμε την πρότασή μα 1η Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε την ενσωμάτωση του κλίματο σε σε όλη την νομοθεσία και είναι ουσιαστική αφορά ειδικά τα ταμεία συνοχής, ε, γεωργίας, έρευνας και ανάπτυξης και την εξωτερική μας πολιτική. Θεωρούμε πως η ενσωμάτωση αυτή πρέπει να είναι ορατή, ευρωστή και όπως τονίζεται από τον οδικό χάρτη του 2050 το να πετύχουμε τους μακροχρόνους στόχους Ένωση περί προσαρμογής σημαίνει σημαντικές επενδύσεις. Βεβαίως, προσθέμενη αξία στον προπολογισμό σημαίνει να εξοδεύσουμε τον προπολογισμό πολύ πιο στοχευμένα σχέση με το που είναι οι πολιτικές μας προτεραιότητες. Π.χ. όταν μιλάμε για ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι σαφές πως θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και περαιτέρω αποτελεσματικότητα και να μειώσει και το κόστος εισαγόμενων ορικτών καυσίμων. Κάτι ακόμα για την περαιτέρω εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Το ένα είναι η ασφάλεια, το άλλο είναι η υποπτία της αγοράς άνθρακα, να περιοριστεί ο κίνδυνος απάτης στο νέο αυτό τομέα και εξετάζουμε επιλογές μεταξύ των οποίων και η κατάταξη αυτών των μέσων ε, στα χρηματοοικονομικά μέσα για να υπαρχούν σχετική οδηγία. Να πω πως δεν εφευρίσκουμε τίποτα το καινούριο προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να τα εντάξουμε σε υπάρχουσες δομές. Για την αεροπορία, δύο διαβάζετε και εφημερίδε. Νομίζω η εφαρμογή της νομοθεσίας για να συμπεριληφθεί η αεροπορία ε, προχωράει. Όλα τα βασικά στοιχεία υπάρχουν ή θα ολοκληρωθούν και μετά θα έχουμε τον ε, δημοσίευση των εναρμονισμένων μέτρων σύγκρισης για άδειες στις αεροπορικές εταιρείες. Πολλά μπορούμε να πούμε, απλά να πούμε πως πρόκειται για μια βασική αρχή που προσπαθούμε εδώ πέρα να περάσουμε και Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν πριν από λίγα χρόνια το έκαναν αυτό λέγοντας πως βεβαίως και η αεροπορία θα πρέπει να συμπεριληφθεί, είναι παγκόσμιο τομέα και βεβαίω δεν μπορεί να αφορά μόνο τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Και οι ανταγωνιστέ του, όταν προσγειώνονται ή απογειώνονται από την Ευρώπη, θα πρέπει να αποτελούν μέρο. Νομίζω πω θα αντιληφθείτε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό από ευρωπαϊκή σκοπιά. Λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πολλά μπορούμε να πούμε από αυτού. Σύντομη θα είμαι. Το Ντέρμπαν φαίνεται δύσκολο για λόγους που καταλαβαίνετε. Έλλειψη προόδου στο Κογκρέσο και αλλού. Αλλά η Ευρώπη προχωράει, σπρώχνει σου μπορεί, για να έχουμε στο δυνατό μεγαλύτερη πρόοδο. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να εφαρμόσουμε όλα όσα συμφωνήθηκαν στο Κανκούν, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ορμή όπως ξέρετε μόνο με την εφαρμογή πρέπει να υπάρχουν και νέα πράγματα αλλά νομίζω πως στην Επιτροπή σας πρέπει να τονίσω πως για να προωθήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις εργαζόμαστε και διμερώς με εταίρους κλειδιά όπως π.χ. η Κίνα για να βρούμε διμερείς ε, συνεργασίες, μηχανισμούς αγοράς με το πώς ρυθμίζουν τα πράγματα στην Κίνα. Θα ξέρετε πως το επόμενο πενταετέ σχέδιο έχουν εδώ πέρα μεγάλα πιλωτικά έργα για το εμπόριο άνθρακα. Το εμπνεύσαμε αυτό και συνεργαζόμαστε με την Κίνα και συνεργαζόμαστε και στην τομιακή συνεργασία μαζί τους και ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κινέζικες ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα έχουμε και εμείς ε, τις βιομηχανίες μας ε, για να ε, έχουμε τους εταίρους μας στην Κίνα. Θα μείνω σε αυτά. Βεβαίως έχουμε και το πρόγραμμα εργασίας κομισιών για του χρόνου, το οποίο προετοιμάζεται με στόχο υιοθέτηση από την Ολομέλεια της Επιτροπής το σώμα στις 26 Οκτωβρίου πέρα λοιπόν από τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές θα δοθεί και άλλη συνέχεια στον οδικό χάρτη του 2050 και επιλογές για το πώς θα πάμε πέρα από τη μείωση του 20% κάτι ακόμα για την αυτιλία. Θα θυμάστε πως πριν από λίγα χρόνια το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Κομισιόν να κάνει κάτι για την αυτιλία. Εάν μέχρι το τέλος του έτους ε, δεν υπάρχει προόδος στον ε, Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να δούμε τι θα κάνουμε στην Ευρώπη. Και εδώ πέρα ο Επίτροπος Κάλλας ε, και εγώ έχουμε ένα φόρουμ των ενδιαφερομένων, συναντιόμαστε τρεις φορές το έτος και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, αν δεν υπάρχει δηλαδή πρόοδος διεθνώς, τι θα γίνει, ποιος είναι ο καλύτερος α, δρόμος να προχωρήσουμε. Θα πάντων ακόμα είμαστε στις διαβουλεύσεις, θα μείνω σε αυτά κύριε Πρόεδρε και μετά οι ερωτήσεις σας θα καθορίσουν το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για την ενημέρωση και σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη βάση για τη συζήτηση και ξεκινάμε με την κυρία Δερκαστήλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι για την ενεργειακή αποδοτικότητα υπάρχει μία προϋπόθεση που καλύπτει όλους τους τομείς τους οποίους ε, συζητάμε. Μειώνονται οι εκπομπές, ενθαρρύνονται η έρευνα και η ανάπτυξη. Ε, πρόκειται για ένα τομέα που μπορεί να έχει πάρα πολύ θετικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς που αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. και θα ήθελα να αναφέρω κάποιες πτυχές που αφορούν τους συγκεκριμένους αυτούς τομείς ε, και συγκεκριμένα την έξυπνη κατανάλωση. Η κατανάλωση, η κατανάλωση ε, μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας, την εξοικονόμηση ενέργειας και ε, επομένως η έξυπνη κατανάλωση που βασίζεται σε έξυπνα δίκτυα και στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης και βασίζεται επίσης και στην επιλογή των καταναλωτών, χρειάζεται πιλωτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, ούτως ώστε να γίνει μια προσαρμογή αυτών των έξυπνων μέσων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσονται τέτοια προγράμματα μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη πολλοί τομείς ε, διαμαρτύρονται ε, για αυτά τα οποία ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα γιατί είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται στις Ηνωμένε Πολιτείε και τα προγράμματα αυτά θα ήταν απαραίτητα. Ε, τι έχει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όλοι αυτοί οι τομείς στους οποίους προανέφερα εμπλέκονται σε τέτοιου είδου προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ούλσκοκ, ευχαριστούμε την Επίτροπο για την εισαγωγική της παρουσίαση. Θα ήθελα, όπως και η συνάδελφός μου, να τονίσω και εγώ ότι τα θέματα ενεργειακής απόδοσης έχουν κέρια σημασία, κυρίως για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Επίσης, καλό είναι να αλλάξουμε γραμμή και να δούμε πού θα κάνουμε τις επενδύσεις μας για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών στις δικές μας χώρες. Ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτό με την επιδότηση για την, ε, τη διεθνή βοήθεια μάλλον για την καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών και να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Τώρα έχουμε περιέλθει στην εξή κατάσταση. Ε, είμαστε μετά το ατύχημα τη Φουκουσίμα και πριν την διάσκεψη του Ντούρμπαν. Μπορούμε να το θεωρήσουμε απειλή, μπορεί να το θεωρήσουμε όμως και ευκαιρία για το μέλλον. Όλοι όσοι συμμετείχαν ε, στην αποστολή των αντιπροσωπιών στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα θα γνωρίζουν, όπως και η Επίτροπος, ότι για να αποσαφινιστεί η εικόνα σε σχέση με τη θέση της Κίνας, γιατί θυμάστε ότι στην Κοπενχάγη ήταν το κακό το παιδί η Κίνα. Στην Κανκούν τώρα η Κίνα είχα, διατηρούσε low profile, ε, ε, ε, κινείται χωρίς να, κάνει, να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες. Αλλά για τον Τούρμπαν ανοίγονται νέες ευκαιρίες μπροστά μας. Δηλαδή μπορούμε να παρακινήσουμε τους ε, Κινέζους να, να δραστηριοποιηθούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και αποκομίσαμε την εντύπωση ότι μας δίνεται αυτή η δυνατότητα την περασμένη εβδομάδα που ήμασταν στην Κίνα. Οπότε σε συνδυασμό με την Κίνα και όχι μόνο και άλλες χώρες θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η διάσκεψη του Ντούρμπαν να είναι γόνιμη γιατί εκπνέει το πρωτόκολλο του Κιώτο και χρειάζεται αντικατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν με μία φωνή και με υψηλέ φιλοδοξίε να κινηθούμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ θα πρέπει να βρούμε κάποιου ισχυρού εταίρου με του οποίου θα συνεργαστούμε για να σημειωθεί η πρόοδο. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ότι δεν θα οδηγήσει σε τίποτα η διάσκεψη του Ντούρμπαν και ότι θα αποτύχουν και θα καταρρεύσουν απογοητεύσουν όλα αυτά που έχουμε κάνει ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ο κίνδυνο ελοχεύει. Είναι πραγματικό. Κυρία Χόλ τώρα. Thank you. Um... Ευχαριστώ την Επίτροπο. Ήταν ε, πληρέστατη η παρουσίασή σας. Μιλήσατε για την ενεργειακή απόδοση και τον κύριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Είπατε ότι αν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα αυτό το θέμα, ε, δεν θα πάμε πουθενά. Μα το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Εγώ ανησυχώ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις βάσει των οποίων η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μπορεί να προσπαθεί να αντιταχθεί στην προσπάθεια υιοθέτηση αυστηρή νομοθεσία για δεσμευτικού στόχου μακροπρόθεσμα. Έτσι, γιατί στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να εκτιμηθεί η δράση των κρατών μελών το 2013, το 2014. Αλλά τελικά η Ένωση τι μπορεί, η Επιτροπή, συγγνώμη, τι μπορεί να κάνει για να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπίσουμε όντω με σοβαρότητα το ζήτημα και το ταχύτερο δυνατόν μάλιστα. Πέραν αυτό υπάρχουν δύο τομεί που ανησυχούν. Η αξιοπιστία των δεσμεύσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητείται και αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό την τελεσίδικη δράση της Επιτροπής. Αυτά τα δύο ζητήματα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Ε, επίσης ε, για την ποιότητα των καυσίμων οι οριακές τιμές ε, ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί επίσης ε, η οδηγία για τη χρήση της ενέργειας. Έχουν σημειωθεί ε, κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Ξέρω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, αλλά θα μας βοηθούσε αν μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Λάμπερτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο. Θα ήθελα να καταδείξω ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ε, κλιματικές αλλαγές και το θέμα που μας απασχολεί σχεδόν από την αρχή της θητεία μας, δηλαδή το θέμα των πόρων. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση για τη χρήση των πόρων, όπου αναφέρεται βασικά ότι αν δεν έχουμε σωστή διαχείριση ούτως ώστε να επιτύχουμε πλήρη αποσύνδεση ανάμεσα στην ε, ανάπτυξη ε, και τη χρήση των πόρων δεν θα εκπληρώσουμε τους ε, κλιματικούς στόχους μας. Ακόμη και είναι η λιγότερο φιλόδεξη μπορούμε να φανταστούμε. Και αφήστε τι θα γίνει μετά το 20%. Δεν το συζητάμε καν. Και ρωτώ το εξή, σα ικανοποιεί πρώτον να μην έχουμε στόχο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ούτε να έχουμε ε, στόχο για την χρήση των πόρων. Αν φτάσουμε ποτέ εκεί, είναι δυνατόν να εκπληρώσουμε τους στόχους μας αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο ε, και με ανησυχεί η στάση της ε, διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα για αυτό το θέμα. Και σε σχέση με το ERP και το IPCC και τα συμπεράσματα του ειδικευμένου πάνελ, δεν θα έπρεπε να προωθεί όχι μέτρα ε, παραγωγής αλλά μέτρησης. Ε, δηλαδή όταν μιλάμε για τη χρήση των πόρων και τους στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα είναι παράλογο να συζητάμε εάν δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι η παραχθήσα ενέργεια στην Κίνα καταναλώνται ουσιαστικά στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Γκέρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και χαίρομαι που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Έχω την εξής ερώτηση. Περισσότερες μάλλον ερωτήσεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα μέτρα τα οποία αναφέρατε. Καταρχήν υπάρχει μία υπόθεση για τις ανθρωπογενείς ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, χωρίς να έχουμε όμως την πλήρη επιστημονική βάση. Ε, υπάρχει άσκηση πιέσεων, ε, μορφής ομάδων πιέσεως, λόμπι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις όμως διότι δεν πρέπει απλώς να απευθυνόμαστε ε, στο ότι πιστεύουμε ότι ε, δεν μπορεί να λέει ψέματα η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Ε, όταν είχα ρωτήσει τον κύριο Δήμα κάποτε μου είχε πει ότι πιστεύει τα αποτελέσματα της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα ακόμη και αν δεν βασίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά αποτελέσματα. το Γεωλογικό Ινστιτούτο στην Πολωνία για την ε, ε, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ε, επαληθεύει τα στοιχεία αυτά και είναι επιστήμονες και η γνώμη τους είναι διαφορετική από τη γνώμη της Επιτροπής. Τρίτον, ο περιορισμός των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες ε, επιστημονικές ανακοινώσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας δείχνουν ότι δεν ισχύουν ε, οι υποθέσεις για ανθρωπογενή αίτια των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. κύριος Γκέμπελς, έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές και θα πρέπει ε, να σας ζητήσω να συντομεύσετε, λέει ο Πρόεδρος ή θα δούμε μήπως να δοθεί μια συνολική απάντηση. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκέμπελς τώρα. Κύριε Επίτροπε, με όλο το σεβασμό που έχω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μερικές φορές νομίζω ότι ε, η Επιτροπή εκφράζεται σαν να πρόκειται για χορό σε αρχαία τραγωδία, ότι όλοι μαζί, ε, ε, ολόκληρη η Επιτροπή εκφράζεται με ενθουσιασμό προτείνοντας να προχωρήσουμε προς τα μπρος ε, και θα ήθελα πάρα πολύ καλά να δω ποια είναι η συγκεκριμένη πολιτική μέχρι το 2020 για να επαληθεύσουμε τους στόχους τους, για να ε, υλοποιήσουμε συγγνώμη, τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά βήματα και ζητάμε και από τις άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν. Εσείς στην Κοπενχάγη ε, σαφώς γνωρίζετε ότι η πρόταση την οποία κάνει η Ευρώπη ε, δεν ενδιαφέρει ολόκληρο τον κόσμο και οι προτάσεις και η συμφωνία της ε, ε, Κοπενχάγης μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει τον πρόεδρο Μπαρόζο, την κυρία Μέρκελ και τον πρόεδρο Σαρκοζή. Και στο Κανκούν παρόμοια αποτελέσματα και το τι θα γίνει στον Τέρμπαν επίσης δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα είναι πολύ θετικό. Είναι γεγονός ότι οι Κινέζοι δεν θα δεχθούν ποτέ ένα σύστημα cap and trade, δεν θα δεχθούν ποτέ το σύστημα του Κιώτο και αφού δεν θα το δεχθούν το σύστημα οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί και οι Ινδοί και οι Βραζιλιάνοι επίσης δεν θα το δεχτούν. Πώς θέλετε λοιπόν να συνεχίζει να δίνει το καλό παράδειγμα η Ευρώπη ενώ οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος ε, μέσα σε πέντε χρόνια από το 14% έχουν περάσει στο 10% των παγκοσμίων εκπομπών δεν μπορούμε να ε, προχωρήσουμε πέρα από τους στόχους μας ανεξάρτητα από ε, το διοξίδιο του άνθρακος. Εγώ νομίζω ότι ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επενδύσουμε κυρίως στην έρευνα, πράγμα το οποίο δεν κάνουμε. Γιατί εδώ υστερούμε σε σχέση με τους Κινέζους και τους Αμερικανούς και πολλούς άλλους όσον αφορά την έρευνα. Σα παρακαλώ λοιπόν ε, κύριε Επίτροπε ότι όλα αυτά το οδικό χάρτη το 2050 και όλα αυτά. Ήδη το είπα στον Επίτροπο Έτσιγκερ. Σα εύχομαι μακροζωία, αλλά λίγοι θα είμαστε το 2050 εδώ για να επαληθεύσουμε το τι θα έχει γίνει με τι προτάσει ε, τη Επιτροπή. Κυρία Καβάλιο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσία της και για τις διεξοδικές ε, διευκρινήσεις της. Χθες ε, ο Γενικός Διευθυντής ε, Προϋπολογισμού μας είπε ότι περίπου 400 εκατομμύρια θα δαπανηθούν για το σχέδιο ανάκαμψης που συνδέεται με το CCS διότι υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή και ένα από τα προγράμματα δεν έχει προχωρήσει. έχετε κάποια πρόθεση να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση, για τα κτίρια, για τις βιώσιμες κοινότητες ή για κάτι άλλο. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, για τις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές μπορείτε να είστε λίγο πιο ε, συγκεκριμένοι. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά ποια νέα στοιχεία προβλέπετε για τον Τέρμπαν ε, κυρίως αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, η διετομιακή συμφωνία δηλαδή με την Κίνα. Πρόκειται για ένα νέο CTM ε, ή θα είστε πιο φιλόδοξοι, δηλαδή στα, ταυτόχρονα με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα ε, προωθήσετε και αυτό, δηλαδή θα έχετε γενικότερους στόχους για ολόκληρη την οικονομία για να αντιμετωπίσετε την διαρροή ε, άνθρακα σε αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους. Σας ευχαριστούμε. Θα απαντήσει η επίτροπο, Έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσεις ε, και γι' αυτό α σταματήσουμε τώρα το γύρο των ερωτήσεων για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Επίτροπο για τι απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν προς την κυρία Ντελκαστήλιο. Μιλήσατε για τα έξυπνα δίκτυα. Ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία επ' αυτού. 80% ε, ε, ε, των οικοκυριών θα πρέπει να έχουν έξυπνους μετρητές μέχρι το 2020. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι και θέματα προϋπολογισμού. Υπάρχουν δυνατότητες μέσω του προϋπολογισμού να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, της έξυπνης υποδομής ενέργειας κλπ. Αυτό συζητάμε τώρα στην Επιτροπή και σίγουρα στον προπολογισμό που θα προτείνουμε μέχρι την 1η Ιουλίου θα φανεί η σημασία που δίνουμε σε αυτές τις προτάσεις και το Κοινοβούλιο ε, επίσης θα έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί για τον προπολογισμό. Προς ε, την Μαρίτα Ουλσκοφ και για το ρόλο της Κίνας ε, εν ώψη των διαπραγματεύσεων στον Τέρμπαν. Όλοι ελπίζουμε ότι είναι μια τέτοια βασική χώρα ε, ε, όπως η Νότια Αφρική θα έχει την προεδρία της ΚΟΠ και επομένως εφόσον μια τόσο σημαντική αναδιόμενη χώρα ε, θα έχει την δυνατότητα να υποβάλει πρωτοβουλίες μπορεί να γίνουν αποδεκτές αυτές οι προτάσεις από πολύ περισσότερες χώρες. Αυτό ελπίζουμε. Είπατε επίσης και εσείς και η κυρία Καρβάλη τι μπορούμε να κάνουμε για τον Τέρμπαν. Υπάρχει ο κίνδυνος οι διαπραγματεύσεις στον Τέρμπαν να μην καταλήξουν σε κανένα από αποτέλεσμα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί για να αποφύγουμε μια τέτοια δυσμενή προοπτική. Γίνεται διάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσα μετά το, το Πάσχα, μέσα στον τελευταίο μήνα, κάναμε ένα φόρουμ μαζί με τους Αμερικανούς και προσπαθούμε ε, να ζητήσουμε από τους ε, επόμενους οικοδεσπότες της ΚΟΠ, τους νοτιοαφρικανούς δηλαδή, να σκεφτούν πιθανά προγράμματα, ε, πιθανά, πιθανές δυνατότητες που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές στο Τέρμπαν. Και μιλάμε για τη δεύτερη περίοδο ε, ε, ανάλυσης δεσμεύσεων, μιλάμε για όλα τα πιθανά προγράμματα. Για να μην αποτύχει όμως το σενάριο αυτό, προσπαθούμε να σκεφτούμε και άλλα πιθανά αποτελέσματα. Πώς να συμπεριλάβουμε την αυτιλία και την αεροπλοεία, πώς να έχουμε συνεργασία, πώς να βελτιώσουμε το σύστημα CDM για τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα συνεχίσουμε και στη Βόνη τον Ιούνιο και με την Νότια Αφρική και τη Γερμανία στις αρχές του Ιουλίου θα προχωρήσουμε επίση προς την ίδια κατεύθυνση για να βάλουμε και άλλα παραδοτέα στη συζήτηση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και μακάρι να είχαμε κάποια θετικά σήματα από την Κίνα όπως ε, αναφέρατε. Η κυρία Χολ ε, ρωτάει αν ε, πραγματικά αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει κάποια έλλειψη λογικής συνέπειας. Ε, οι επιχειρηματίες με τους οποίους συζητώ και όλες οι κυβερνήσεις ε, έχουν να πούνε ότι ε, όλα αυτά είναι λογικά και η οικονομική λογική υπάρχει πίσω από αυτά, αλλά δεν βλέπουμε να προχωρεί σημαντικά το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και γι' αυτό το πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας που παρουσίασε ο Επίτροπος Έτιγκερ και μέρους της Επιτροπής περιλαμβάνει κάποιες ριζικές πρωτοβουλίες, όπως παραδείγματος χάρη ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει κάθε χρόνο να φροντίζει για το 3% των δημοσίων κτηρίων σε ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, εγκαθιστώντα σε υφιστάμενα κτίρια τα κατάλληλα συστήματα για ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα χρειαστούμε ε, λοιπόν ε, και κονδύλια μέσω του προπολογισμού για να προωθήσουμε καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότηση και είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνούμε. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένα κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη, νέα κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη, έχουν αρχίσει να εξετάζουν το θέμα τη ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί βλέπουν ότι είναι κάτι που βολεύει την οικονομία του θα γίνει μια διαβούλευση την Παρασκευή ε, ε, ακριβώς για θέματα ε, ενεργειακής αποδοτικότητας και έχει κληθεί να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετά δύσκολα θέματα. Ε, τώρα έχουν δοθεί προς αξιολόγηση από τους ομοτήμους για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις ως επόμενο βήμα σε αυτόν τον τομέα. Σε σχέση με τι ερωτήσει του κυρίου Λάμπερτ, νομίζω ότι γενικά απάντησα όσον αφορά του στόχου ενεργειακή αποδοτικότητα, και αν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Για το αν πρέπει να έχουμε και ένα στόχο για αποδοτικότητα των πόρων, για πρώτη φορά φέτο θα υποβάλει η Επιτροπή μια ανακοίνωση για την αποδοτικότητα των πόρων. Και συμφωνώ μαζί σα, κατά βάση ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και γι' αυτό είναι και εμβληματική μα πρωτοβουλία αυτό. και τα μέτρα τα οποία αφορούν ε, την παραγωγή ε, είναι μέτρα στα οποία θα ήθελα να σας παραπέμψω στην οδηγία για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε φορολογικά έσοδα στην ε, Ευρώπη ε, μέσω της φορολόγησης της εργασίας, αυτό θα βλάψει την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα μας, ωφελούσε, θα μας αν ε, φορολογούμε την κατανάλωση των ενεργειακών πόρων και όχι την, να φορολογούμε την εργασία. Αυτό είναι, αυτή είναι μία από τις πιθανές οδούς που διερευνούμε και με τον κύριο Γκίρεκ ε, δεν, ε, δεν ξέρω τι έχω να σας πω για τα σχόλιά σας, αν σωστά σας κατάλαβα. Τονίσατε τις ε, ανθρωπογενείς, τα ανθρωπογενή αίτια. Ίσως δεν υπάρχουν απόλυτα τεκμηριωμένα συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι και όσοι δεν πιστεύουν ότι ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι βλέπουν ότι υπάρχει ε, λόγος ε, να υποστηρίξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί τουλάχιστον επενδύουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία και όχι σε χώρες εκτός Ευρώπης για μη αποδοτικές επενδύσεις και πιστεύω ότι μειώνουμε ε, τις εκπομπές ε, απαντώντας τον κύριο Γκέμπελς. Διαφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι δεν ε, θα δεχθεί η Κίνα το σύστημα Cap and Trade. Δεν έχετε δίκιο γιατί ήδη το κάνουν τώρα σε έξι πιλωτικά προγράμματα. Στη Σανγκάη, το Τσάνγκ τη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, στο Πεκίνο, στο Τσίνγκ στο Γουαντόγκ, σε βασικές βιομηχανικές πόλεις το 2012 και 2013 προσπαθούν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, αυτούς τους μηχανισμούς του ε, cap and trade. Και το ανέφερε και ο Κινέζος Υπουργός ότι δεν αρκεί να θέτουμε στόχους. Θα πρέπει να τους ε, ε, επιδιώκουμε χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς της αγοράς. Θέλω να πω ότι προχωρούν και εκείνοι και προσπαθούμε εμείς διμερώς μαζί τους ε, ούτως ώστε το σύστημα που θα εφαρμόσουν οι Κινέζοι να είναι κατά κάποιο τρόπο συγκρίσιμο με το σύστημα που έχουμε και εμεί στην Ευρώπη. Και για τι ε, διαρροέ διοξιδίου του άνθρακα ε, καταλαβαίνω του φόβου που έχετε και γι' αυτό ε, προσπαθούμε μέσω benchmarking να δούμε ποιοι είναι οι τομεί στου οποίου μπορούμε κυρίω να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μα. Αλλά και οι ανταγωνιστέ μα κινούνται προ αυτήν την κατεύθυνση και δεν πρέπει να υποτιμούμε τι προσπάθειές του. Συμφωνώ μαζί σα ότι στον επόμενο προπολογισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη. Η καινοτομία θα είναι το κλειδί για την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μπορούν να συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να δοθούν νέε προτεραιότητε στο νέο προπολογισμό σε σχέση με του παλαιού προπολογισμού. Διαφορετικά, τελικά δεν θα έχουμε αρκετού πόρου για να κάνουμε αυτά τα οποία καλύτερα θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, μαζί. Αυτά προ το παρόν. Ε, τέθηκε ένα ερώτημα για τα 400 εκατομμύρια σχετικά με το πρόγραμμα ανάκτηση. Δεν ξέρω ακριβώ ε, πού πηγαίνουν αυτοί οι πόροι, αλλά μετά τη συνεδρία, κυρία Καρβάλιο, θα μπορούσα να επανέλθω σε αυτό το θέμα να σα δώσω στοιχεία. Um Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρέμβαση. Συνήθω δεν παρεμβαίνω, αλλά θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη ε, παρέμβαση για τον κύριο Γκέμπελ. Ευχαριστώ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την Κίνα και ε, σε μια πενταετή περίοδο πήγαινα συχνά στη Σανγκάη για ε, την, παγκόσμια εκθέση. Λοιπόν, η Σανγκάη έχει ως στόχο μέχρι το 2020 να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Και θα το καταφέρουν γιατί επενδύουν. Ενώ εμείς μιλάμε, δεν επενδύουμε. Και αυτό καταγγέλλω εδώ. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε και έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε υπόψη. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω μόνο και να κλείσω έτσι. Η Φουκουσίμα οδήγησε στο ότι δεν συζητάμε μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο περί τεστ αντοχής ε, πυρηνικών εργοστασίων κτλ. αλλά και σε κάποιες χώρες, δηλαδή στη δική μου, στη Γερμανία, μιλάμε για μία, έναν ε, αναπροσανατολισμό και μάλιστα απομάκρυνση από την πυρηνική ενέργεια μέχρι το 2020-2025. Αυτό οδηγεί στο ότι ε, σκεφτόμαστε πώς θα υποκαταστήσουμε την πυρηνική ενέργεια και αυτό οδηγεί στο ότι βεβαίω θα επεκταθούν οι ανανεώσιμες πηγές αλλά και στον τομέα των υπολείπων θα μιλήσουμε για άνθρακα, και υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο και θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις για να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και δεν μιλάμε πια τόσο πολύ για την προστασία του κλίματος σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια Οπότε οδηγεί στο ότι όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι ε, αμφισβητούνται πάλι. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, χθε είχαμε τους συναδέλφους εδώ πέρα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και διήθυνε ο πρόεδρος ε, την συζήτηση και υπενθύμησαν κάποιοι πως όχι μόνο στη Γερμανία αλλά γενικώ παγκοσμίω ε, θα αυξηθεί η ζήτηση αερίου Εν ολίγης δηλαδή έχουμε εξελίξεις ε, τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες που αμφισβητούν ε, τους ε, στόχους μας. ε, Βεβαίως εγώ είμαι υπέρ του πακέτου που εγκρίναμε το 2008 τότε είχαμε βεβαίως τον τότε πρόεδρο, αλλά το πώς θα έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους χωρίς να βλάψουμε ε, την ανταγωνιστικότητά μας και να οδηγηθούμε σε αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης είναι κάτι που με ανισχύει. Εγώ φοβάμαι μια σταδιακή αποβιομηχάνηση της Ευρώπης. Βλέπω ο πρόεδρο κοιτάει το ρολόι. Κοιτάξτε, έχουμε τεράστια προβλήματα με τη σταθερότητα του ευρώ. Έχουμε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, έχουν ακριβώς μεγάλα προβλήματα γιατί δεν είχαν καθόλου βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα, για να το πω απλά, ε, θέλουμε κάποια στιγμή να της δώσουμε την ευκαιρία να σταθεροποιηθεί. Ε, ξέρετε πως υπάρχει μια συζήτηση περί ενός σχεδίου Μάρσαλ και πως θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία, όποια βιομηχανία και αν είναι. Εντάξει θα υπάρχουν και πράσινες βιομηχανίες, αλλά εάν μιλάμε για βιομηχανία θα έχουμε πάλι επιβάρυνση του κλίματος και Ξέρω πως η αποστολή σας είναι άλλη, εσείς είστε η Επίτροπος Προστασίας του Κλίματος στην Ευρώπη και τα λοιπά, Αλλά σας παρακαλώ να μην γίνει αυτό εις βάρος της βιομηχανίας μας. Εάν γίνει αυτό και φύγουν οι βιομηχανίες και οι θέσεις εργασίας στην Κίνα και στον αραβικό χώρο και οπουδήποτε αλλού, ε, να αναφέρω π.χ. μόνο ως παράδειγμα τη χημική βιομηχανία, αν δείτε τι γίνεται στο Κατάρ από ευρωπαϊκές εταιρείες, τότε φοβάμαι πάρα πολύ και δεν ξέρω Ελπίζω να ακολουθήσετε τη σωστή πολιτική πορεία. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ κοίταξα το ρολόι ε, για το ότι έχουμε μόνο άλλα 15 λεπτά. Οπωσδήποτε χρειάζεται 5 λεπτά η κυρία Επίτροπης για να απαντήσει. Έχουμε 10 λεπτά και 6 ακόμα μιλητές, οπότε υπολογίστε τα μόνοι σας. Ο κύριος Ζαντό. Δεν είμαι πολύ καλός στους υπολογισμούς, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, Euh, πρώτο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω, πρώτη ερώτηση μάλλον. Ε, κατά τη γνώμη σας, ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, της έκθεσης των εκθέσεων που ψηφίστηκαν και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την κατάσταση μετά το 2020. Και πάλι περνάει ένα ηχηρό μήνυμα το Κοινοβούλιο, πιέζει στην Ευρώπη να κάνει περισσότερα πράγματα, να τα κάνει καλύτερα και όχι μόνη της. Γιατί ο στόχος είναι να έχουμε μια δυναμική, αλλά να αναλάβουμε και ηγετική θέση στην παγκόσμια μια σκηνή. Δεύτερη ερώτηση. Πού βρισκόμαστε ε, για τις ε, χρηματοπιστωτικέ δεσμεύσεις των χωρών ΩΣΑ και κυρίως ε, των ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια των μηχανισμών που θεσπίστηκαν στην Κοπενχάγη και επιβεβαιώθηκαν στην Κανκούν. Και τρίτη ερώτηση. Χθε στην Επιτροπή Ίντα ερώτησα τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για το θέμα μας με τη Μαλαισία τους ε, ρώτησα στις εμπεροκές διαπραγματεύσεις ε, που συνεχίζονται τώρα με την Μαλαισία πέρα από το να υπενθυμίζουμε τα κριτήρια βιωσιμότητας για την εκμετάλλευση ε, του φινικέλαιου θα, δεν θα έπρεπε να αναφερθούμε εξ σε όλες τις γης που αγοράζει η Μαλαισία τώρα στην Αφρικανική Ήπειρο και άρα συμμετέχει στην απερίμωση και την θέρμανση του πλανήτη και μου έδωθη μία απάντηση που θα τη χαρακτήριζα τουλάχιστον αμφίσιμη. Έχετε άλλες πληροφορίες εσείς. Ο κύριος Σώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις και απευθύνομαι ε, στο συνάδελφο Δέλφο Γκέμπελ, αλλά βλέπω ότι φεύγει. Η παρουσία του Νίκολα Σαρκοζή και της Άγγελα Μέρκελ ε, ε, ορισμένες δεν ξέρουμε Ορισμένες φορές είναι καλύτερα να είναι παρόντε ή όχι. Και δεύτερη ερώτηση, ε, έχουμε μία διαφορά με την Κίνα. Η Κίνα δεν είναι δημοκρατία και φυσιολογικό είναι σε ένα δημοκρατικό... Σε, όταν ε, λειτουργούμε μέσα σε μία δημοκρατία να έχουμε μεγαλύτερες συζητήσει. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην οποία ε, βρίσκεστε. Το αναγνωρίζουμε λόγω τη νέα εντολή. Α, και γι' αυτό που έλεγε ο συνάδελφο για τη Μαλαισία. Ε, θα ήθελα περισσότερε πληροφορίε ή δυνατόν για την εμπορική πολιτική τη Ένωση και συγκεκριμένα την εισαγωγή ε, περιβαλλοντικών ρητρών μέσα στι εμπορικέ συμφωνίε. Από πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα το ζητάμε αυτό. Έχουμε πλέον όμω το δικαίωμα, όπω και η Αμερικανική Γερουσία, τηρουμένων των αναλογιών, να εμποδίζουμε την υπογραφή τέτοιων εμπορικών συμφωνιών. Ε, την περασμένη εβδομάδα όταν ε, ε, μιλούσαμε για τις διαπραγματεύσεις του Μερκοσούρ επ' της αποστολής στην Ουρουάη μας είπαν ότι αν επιδιώκεται ΠΟΕ ΣΥΝ δεν θα μπορεί να εισαγάγετε τέτοιε περιβαλλοντικές ρήτρε, γιατί αυτό το απαγορεύει ο ΠΟΕ αλλά περιβαλλοντικές, αμυγός περιβαλλοντικές και διατάξεις ε, για την ασφάλεια μπορείτε να τις συμπεριλάβετε. Οπότε στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε μπορούμε να επιδιώξουμε τουλάχιστον αυτό, κύριος Φλόρενς. Ε, κύριος Φλόρενς. Ε, κύριε Επίτροπε, εγώ 20 χρόνια πάω σε κλιματικές διασκέψεις και απορώ που πάλι σήμερα έχουμε τη συζήτηση για τους αριθμούς και όλοι θεωρούν πως είναι τόσο αποφασιστική στο Τέρμπαν το θέμα είναι ένα. Θα έχουμε μία συνθήκη ή όχι. Και εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε βάρος. Η συζήτηση χτες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος καλή ήτανε, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός των αριθμών δεν οδηγεί πουθενά. Απαριθμούμε συνέχεια τι κάνουν οι Κινέζοι και τι κάνουν οι λοιποί. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε ένα νέο κατάλογο και να προσπαθήσουμε να τα επιτύχουμε βεβαίως. Θα χρειαζόταν και μια μελέτη την οποία αναφέρατε. Α, βεβαίως αυτό έρχεται από το Συμβούλιο, δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το βάρος του 20% που συμφωνώ ανεπιφύλακτα και με το 30% εάν ακολουθήσουν και άλλοι. Αλλά ποιο είναι το κόστος εδώ πέρα. Γιατί στη χώρα μου στη Γερμανία θα πρέπει να ξέρετε πως είναι θέμα να το αποδεχτούν αυτό. Οπότε υπάρχει αυτή η μελέτη και για την απόφαση της, ε, της Ιαπωνίας. Κοιτάξτε, πρέπει να το απαντήσουμε αυτό και μια πραγματική επιθυμία. Γράψτε κάπου τι κάνουν οι άλλοι χωρίς να υπογράφουν ε, συνθήκες και να πω στον κύριο Γκίρεκ δώσω αν δεν είναι αυτή η δική μου φιλοσοφία εγώ είμαι στο πλευρό της κυρίας Νίμπλερ αλλά πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα γιατί κάνουμε αυτές τις μεγάλες προσπάθειες στην Ευρώπη. Ε, τι κάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε όλοι υπεπισμένοι ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα ήθελα κυρίως να μιλήσω για τον τομέα των κτηρίων, γιατί είμαι εισηγήτρια για την οδηγία αυτή και θα ήθελα μέσα στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη 4% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Δεν είναι υποχρεωτικός όρος, αλλά θα πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση σε μια τέτοια δυνατότητα. Ο κ. Ζαντό μίλησε για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες ε, ήταν οι εκπομπές τη δεκαετία του 90 και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μείωσε η Ρουμανία τις εκπομπές της σε σχέση με το επίπεδο της δεκαετίας του 90 κατά 40% το 2005 και αυτό όχι διότι η παραγωγή μας έχει γίνει αποτελεσματικότερη αλλά έγινε αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, έκλεισαν κάποιες επιχειρήσεις, μείωσε επομένως, ε, μειώθηκε το δυναμικό και έτσι μειώθηκαν οι εκπομπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίναμε περισσότερο αποδοτικοί και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που είπε η κυρία Νίμπλε, ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να λειτουργούμε με τρόπο περισσότερο οικολογικό και αποτελεσματικό και όχι να μειώνουμε την βιομηχανική μας ε, δυνατότητα γιατί έτσι θα χάσουμε απασχόληση. Όσον αφορά την χρηματοδότηση δεν μπορούμε να θέτουμε υποχρεωτικού στόχου για μείωση των εκπομπών χωρίς να χρηματοδοτούνται τα απαραίτητα μέτρα και δυστυχώ στον Ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν υπάρχουν τέτοιες ε, εναλλακτικέ λύσεις, δεν δίδονται κονδύλια για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ή των βιομηχανικών κλάδων ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί. Τέλο, κύριε Επιτρόπε, μια τελευταία παρατηρήση όσον αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων εκπομπών υπήρξαν προβλήματα και γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει και απάτες όσον αφορά το ΦΠΑ και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προβλέπετε για να γίνει λειτουργικό αυτό το σύστημα και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Γόντε. Ευχαριστώ. Ίσως είναι κάπως προκλητική η ερώτησή μου. Αλλά με γνωρίζετε, Επίτροπε, και νομίζω ότι θα δεχτείτε την ερώτησή μου. Πραγματικά πιστεύετε ότι η πορεία των Ηνωμένων Εθνών είναι η σωστή πορεία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι το Κανκούν ήταν σαν να προσπαθούσαμε να ξαναδώσουμε ζωή σε έναν σχεδόν νεκρό φορέα. Δεν λέω ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, αλλά γενικά μια τέτοια εικόνα υπάρχει. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ κατά Νομίζω ότι θα είχε νόημα ε, να περάσουμε σε ένα εντελώς νέο προβληματισμό του όλου πλαισίου χωρίς αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ. Ε, μιλήσατε για τον Τέρμπαν ε, που θα λάβει η χώρα επί Πολυνικής Προεδρίας ε, και θέλω να σας ρωτήσω ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος ιδανικά αυτής της χώρας. Ε, θα, θα ήθελα κατά τη διάρκεια της Πολωνικής ε, Προεδρίας να αλλάξει η στάση μας. Θα ήθελα να προχωρήσουμε, να περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό που μας έλεγε η συνάδελφος Νίμπλερ, ε, όντως πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στον, στην ανταγωνιστικότητα και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν χρησιμοποιήσουμε, ή μάλλον, ε, αν δεν χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια, τότε θα πρέπει να στραφούμε προς το φυσικό αέριο. Τι πιστεύετε για το φυσικό αέριο σχιστολίθου και τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην Πολωνία και σε άλλα μέρη της ε, Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα την ε, κυρία Επίτροπο. Είναι πολύ δύσκολο το καθήκον που σας αναθέσαμε. Τέλος πάντων, απαντήστε σε ό,τι μπορείτε. Ευχαριστώ προς την κυρία Νίμπλερ γιατί θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως, είναι, όπως ε, είπατε είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να υστερήσουμε ως προς την ανταγωνιστικότητά μας. Όλοι θα συμφωνήσουν γι' αυτό. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την άσκηση σύγκρισης, benchmarking με τα ορόσημα, για, να, για τους, ε, να δούμε ποιοι είναι οι πλέον εκτεθειμένοι τομείς ε, εκτός Ευρώπης, ε, ποια είναι τα ενεργειακά τους κίνητρα, γιατί πρέπει να δοθούν δικαιώματα δωρεάν σε αυτές τις εταιρείες. Τώρα για την απόδοση, για την εξοικονόμηση ενέργειας, προφανώς είναι βασική μας γραμμή και αυτό είναι ένα από τα διδάγματα από την Ιαπωνία. Ο Πρωθυπουργός κάνει ήδη χτες το είπε και σήμερα νομίζω θα το ακούσουμε και από την G8. Ε, ένα από τα διδάγματα αυτό ήταν ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και εξοικονόμηση, εξοικονόμηση, εξοικονόμηση. Και μιλάνε, μιλάμε για την πιο αποτελεσματική ε, χώρα του κόσμου ως προς την ενεργειακή απόδοση, την Ιαπωνία και αν είμαστε κι εμείς έξυπνοι, αν παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας θα τονώσουμε την καινοτομία τι δημιουργικότητά μας και θα ενισχυθεί η θέση μας ε, στις αγορές όπου ξέρουμε ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα η αύξηση τα προσεχή έτη. Ε, αυτό δεν ισχύει για όλες τις αγορές, αλλά ε, οι αγορές ε, για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακά αποδοτικά θα γνωρίσουν πολύ σημαντική αύξηση της ζήτησης. Όποια μελέτη, όποια ανάλυση και αν δείτε συμφωνεί. Θα τριπλασιαστεί η ζήτηση μέχρι το 2020 και άρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που έχουμε. Να κατάλαβα καλά τα σημάδια της γερμανικής κυβέρνησης, αυτό σκέφτονται ακριβώς. Δηλαδή να δημιουργήσουν θέσεις που θα τονώσουν υπονομεύσουν όμω ε, την ανάπτυξη στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Όχι το αντίθετο, όχι να υπονομεύσουν την ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται ευφυή χειρισμό. Ε, Εσεί με ρωτήσατε για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώ ε, χρήσιμη είναι. και κυρίως αν σε κάθε κράτος μέλος εξεταστεί προσεκτικά για να διαπιστώσουν τις αδυναμίες τους ε, τα κράτη-μέλη προς το παρόν. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια συνεργάζονται με αποφασιστικότητα προσπαθώντας να πιέσουν προς τη σωστή τη λογική κατεύθυνση και πιστεύω ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, δίνει έμφαση σε αυτό. Ε, τώρα για την Αφρική, για το Φινικέλαιο, κοιτάξτε... Υπάρχει το θέμα της ε, αναδιανομής της γης ε, στην Αφρική και θα μας απασχολήσει ε, τα προσεχή χρόνια και εάν συνεχίσει να αυξάνεται η τιμή κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα από τους βασικότερους λόγους γιατί ε, μέσως αλλάζει η χρήση της γη, δηλαδή. εάν δεν κάνουμε σωστέ κινήσει για τα βιοκαύσιμα, τότε θα δημιουργήσουμε σοβαρά προβλήματα επισητιστικά ε, στην παραγωγή τροφίμων. Και γι' αυτό σα μιλούσα για τα κριτήρια βιωσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία του. Ε, ε, Επίση, μα είπατε για τη συμπερίληψη, κύριε Οντή, στι εμπορικέ συμφωνίε περιβαλλοντικών κριτηρίων. Για τον Μέρκοσουρ είναι σαφή η απόφαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το συζητήσαμε πέρσι. Οπωσδήποτε πρέπει να επιδιώξουμε αυτό το στόχο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τον Μέρκοσουρ. Αυτή είναι η στάση τη Επιτροπή. Φλόρενς για την επίτευξη συμφωνίας ή όχι στον Τέρμπαν, τι κάνουν οι Κινέζοι κτλ. Λοιπόν, για τη διαφάνεια και το MRV και για την παρακολούθηση. Ε, νομίζω ότι ε, δεν έχουμε ε, εξίσου καλά αποτελέσματα όσο αναμέναμε και είδατε ότι στην προηγούμενη δέσμευση της Κοπενχάγης, δηλαδή είδατε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στην Κανκούν. Τώρα αν θα έχουμε δεσμευτικές συμφωνίες, όχι δεν νομίζω, όχι επειδή θέλει η Ευρώπη, επειδή άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν το θέλουν. Και γιατί να μην εγκαταλείψουμε αυτή τη διαδικασία όπως ισχυρίζονται κάποιοι ε, θα σας υπενθυμίσω κάτι. Ε, πριν από τρία χρόνια, όταν βγήκε το ενεργειακό πακέτο, η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή του κόσμου, πέρα από την Νορβηγία και την ε, ε, Ελβετία που ε, ήμασταν οι μόνοι που θέσαμε στόχους. Σήμερα πάνω από 90 χώρες έχουν προσυπογράψει τη Συμφωνία Κοπενχάγης και έφεσαν ε, βάσει αυτής της συμφωνίας στόχους. Δηλαδή το έγγραφο που προέκυψε μετά την Κανκούν. Δεν είναι εξίσου φιλόδοξα όσο θα θέλαμε αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν αλλάξουν άλλες μεταβλητές, μπορώ να σας πω ότι εξυπηρετούνται τα επιχειρησιακά συμφέροντα, επιχειρηματικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι χώρες G20 εκτός από τη Σαουδική Αραβία έχουν εγχώριους στόχους. Πολλοί δεν θα θέσουν διεθνώς δεσμευτικούς στόχους, αλλά θα τους προωθήσουν μέσα από την εσωτερική τους νομοθεσία. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει για το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Και στην Κορέα το κάνουν τώρα και ε, σε διάφορα προγράμματα στην Κίνα, η ΕΕ, η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, η Καλιφόρνια τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυση ε, τέτοιου συστήματο. Βέβαια δεν προχωρούν με ικανοποιητικού ρυθμού, πόρο απέχουν, αλλά προ τα εκεί πιέζουμε και στο τέλο ποιο έχει τα μεγαλύτερα συμφέροντα, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Γιατί ε, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι προ συμφέρον των επιχειρήσεων επιχειρήσεων να έχουμε ένα διεθνέ πλαίσιο και όχι μία εκατοντάδα διαφορετικών συστημάτων ε, ε, βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν. Δεν λέω ότι θα πρέπει όλα τα αυγά μα να τα ρίξουμε στο ίδιο καλάθι σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, ε, να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο ή να καταλήξουμε σε αδιέξοδο. Αλλά θα συνεχίσουμε και τη διμερή συνεργασία με την Κίνα, με την Ινδία, με την Καλιφόρνια, με άλλε ισχυρέ οικονομίε. Δεν έχουμε μονομανία και ασχολούμαστε δεν ασχολούμαστε μόνο με τι διεθνεί διαπραγματεύσεις. Ο Φλόρεν με ρώτησε τι κάνει η Ιαπωνία. Ο Καν ναι, θα, θα το πει. Νομίζω ότι οι διεθνώς δεν πλήρουν ε, τις υποχρεώσεις τους. Χρειάζεται ένα νέος βιώσιμος τρόπος ε, διαχείρισης κατάστασης γιατί είδαν ποια, είναι, ποια δυνατότητα έχει η βιομηχανία να αναλάβει ηγετικό ρόλο με το ατύχημα. Μία από τι μεγαλύτερε αλλαγέ που είδαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημοσίευση πέρσι το Μάιο τη ανακοίνωση είδαμε αν προχωρήσουμε προς το 30% ποια θα, θα είναι τα ωφέλη, ποιο θα είναι το κόστος κτλ. Τώρα, σήμερα βλέπουμε ότι καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συζητείτε το θέμα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αντί να είμαστε κοντόφθαλμοι και να προετοιμάζουμε επιμέρου πολιτικέ, ε, εξετάζουμε το πώ με ευφυή τρόπο θα χειριστούμε την κατάσταση για να ε, βοηθηθούν και οι ανταγωνιστέ μα, ε, όχι για να του υπονομεύσουμε. Αυτό σημαίνει, Πρόεδρε, ότι δεν έχουμε σταυρώσει τα χέρια και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι για να ακολουθήσουμε. Διότι θα χρειαστεί χρόνος ε, προτού αναλάβουν δεσμεύσεις ε, στην Τράπεζα ε, των Διεθνών Διαπραγματεύσεων. Αλλά ας μην ε, ξεχνούμε ότι παρότι στις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν, σημειώνουν πρόοδο ε, εγχωρίως στην εθνική τους οικονομία και έτσι δεν πρέπει να συνεχίσουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτές τις αγορές. Και ένα τελευταίο να σας πω, επιτρέψτε μου, πριν από δύο μέρες Πήγα να δω αυτό το αεροσκάφος ε, που ε, βρίσκεται τώρα ε, στο Ζάβεντεμ που κινείται μόνο με ηλιακή ενέργεια, με παλμούς και μοιάζει με Airbus που πέταγε 26 ώρες σε συναπτές χωρίς καμία στάση χάρη στους ηλιακούς συλλέκτες που έχει πάνω του το αεροσκάφος. Δεν είναι το, το πιο ενδιαφέρον πράγμα δεν είναι ακριβώς ότι κινείται με την ηλιακή ενέργεια αυτό το αεροσκάφος. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν 18 χορηγούς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης για, την, ε, για το project αυτό. Να ένα αυτό ζωντανό παράδειγμα πώς αν το επιθυμείτε μπορείτε να ε, χρησιμοποιήσετε τεχνολογίες, εχμής τεχνολογίες κλειδιά που μπορείτε να ε, τις χρησιμοποιήσετε στη χημική βιομηχανία σε διάφορε βιομηχανίε, βιομηχανίες, όπως νέα υλικά παραδείγματος χάρη. Ε, αυτό το σκάφος ζυγίζει ως ένα αμάξι, είναι απίστευτο. Ε, ποιο είναι το μήνυμα αυτών των εταιριών των χορηγών ε, που πήρα πριν από δύο χρόνια. Σε παρακαλούμε Ευρώπη λένε ε, μην καθυστερείς άλλο. Έχουμε την ευρηματικότητα, την την παραγωγικότητα αλλά από την πλευρά σας εσείς πολιτικοί πρέπει να είστε φιλόδοξοι και μακρόπνοες προβλέψεις να μας δίνετε, να κάνετε τις επενδύσεις για την έρευνα. Δεν έχουμε χάσει ακόμη το παιχνίδι. Μπορούμε να είμαστε σε, ε, αλλά χρειάζεται ε, κίνητρο, παρακίνηση. Να ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να κατακτήσουμε τις αγορές και να χρησιμοποιήσουμε ω κινητήριο δύναμη την προσπάθεια που κάνουμε για τις κλιματικές αλλαγές στον τομέα της βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για το πόσο είστε ενδιαφέρεστε αυτό το θέμα. Λοιπόν, διακόπτη συνεδρία, τα λέμε σε κανένα δυο ώρες.